Okay, good afternoon everybody. Um... Καλησπέρα σας. Μου φαίνεται λίγο περίεργο που κάθομαι εδώ, γιατί συνήθως είμαι από την άλλη πλευρά. Αλλά σήμερα είναι ιδιαίτερα με, ε, ιδιαίτερη μέρα, γιατί κανένας από τους προέδρους και αντιπροέδρους δεν είναι διαθέσιμος για τη σημερινή συνεδρίαση. Ελπίζω βέβαια στη διάρκεια της συνεδρίασης να έρθει και κανένας συνάδελφος. για την ημερήσια διάταξη να σας ενημερώσω ότι το σημείο 6 πώληση ηθαγένεια στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκή Ένωσης και καταγγελίες περί διαφθοράς ε, στην έκδοση τίτλων διαμονής και θεωρήσεων από προξενία και πρεσβείες κρατών μελών σε τρίτες χώρες και συνέπειες για την ασφάλεια της Ένωσης, αναβάλλεται για άλλη συνεδρίαση. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις λοιπόν, Εγκρίνεται η μερίσια διάταξη. Δεύτερον, δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχει διερμηνία σε, στα Ιρλανδικά, στα ε, Δανέζικα και στα Κροατικά. Και μια τελευταία ανακοίνωση. Οι ψηφοφορίες θα γίνουν στις 6 και 20 σήμερα. Ναι. Καλό είναι να έχετε όλες τις κάρτες ψηφοφορίας σας λοιπόν για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε το συντομότερο δυνατόν και χωρίς προβλήματα. Έχουμε κάτι κρεμότητες για την έγκριση των πρακτικών. Έχουμε τα πρακτικά της 30ης Μαρτίου μέχρι και 1η Απριλίου 2015, 28-29 Μαΐου 2015 και τη συνεδρίαση της Δευτέρας Ιουλίου 2015. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις για τα πρακτικά, θεωρούμε ότι εγκρίνονται. Ωραία. Συνάδελφοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε τώρα με το πρώτο ουσιαστικό σημείο στην ημερήσια διάταξη, το σημείο 4, νομική συνδρομή για ή κατηγορουμένους που στερούνται την ελευθερία τους και τη νομική συνδρομή σε διαδικασίες εκτέλεσης του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Θα Ακούσουμε σήμερα πώς έχουν οι διαπραγματεύσεις ε, σε τριμερές επίπεδο για αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα για τις ε, δικαστικές διαδικασίες. Πρόκειται για το σχέδιο οδηγίας, όπως σας είπα, για την ε, νομική συνδρομή για υπόπτους κατηγορημένους που στερούνται την ελευθερία τους και τη νομική συνδραμή σε διαδικασίες εκτέλεσης του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Θα δώσουμε πρώτα το λόγο στον εισηγητή, στον Τένις Ντεγιόν, για να μας παρουσιάσει πώς έχει κατάσταση και μετά θα δώσουμε το λόγο στους υπόλοιπους συναδέλφους. Ντένις. Uh, um, um, Σε ευχαριστώ, Πρόεδρε, και νομίζω το γεγονό ότι κανεί δεν είναι εδώ είναι καλό σημάδι, καλή ένδειξη. Γιατί σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αμφιλεγόμενα σημεία. Με αυτό το πνεύμα, λοιπόν, κινούμαστε από την αρχή του έτου. Στην τελευταία παρουσίαση είπαμε στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ότι δεν είχε σημειωθεί τότε ουσιαστική πρόοδο ε, με την προηγούμενη Προεδρία, αλλά ήταν αρκετά επικοδομητική αυτή η τελευταία περίοδος, γιατί εξετάσαμε τα επιχειρήματα του ένας του άλλου, προσπαθούμε να δείξουμε μια κατανόηση και νομίζω ότι υπήρχε καλή πρόθεση και από την Ολλανδική Προεδρία και από τη δική μου πλευρά για να δούμε μήπως μπορούσαμε να ακολουθήσουμε μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση. Να μην καταλήξουμε σε μια κατάσταση ιδεολογικού αδιέξοδου, στην οποία δεν θα μπορούσαμε να σημειώσουμε καμία πρόοδο και σίγουρα και λόγω της ε, και χάρη στην ε, Προεδρία του Λουξεμβούργου καταφέραμε φέτος να ξεκινήσουμε με το διδακτικό, με τα ίδια άρθρα και σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό ένταλμα, το άρθρο 5 μας φαίνεται ότι θα είναι δυνατόν να πετύχουμε συμφωνία για το άρθρο 5 παρά για τα άλλα άρθρα συζητήσαμε και το άρθρο για την ποιότητα της νομικής αρρωγής σε ό,τι αφορά τα όσα είχαν παρουσιαστεί και προηγουμένως ε, στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θεωρούμε ως Κοινοβούλιο ότι σημαντικό θα είναι να αποτυπώνονται κάπως και τα, το περιεχόμενο της οδηγίας. Έχουμε λοιπόν κανονίσει και άλλες συναντήσεις, άλλες τέσσερις με την Ολλανδική Προεδρία. Θεωρώ ότι μπορούμε να πούμε ότι έχει συμβιωθεί πραγματικά πολύ πρόοδο σε ό,τι αφορά το άρθρο 5. Και στο 5α όμως, όπως ονομάζεται πλέον το κεφάλαιο που είναι αφιερωμένο στην ποιότητα της νομικής αρρωγής, υπάρχουν κάποιες διαφορές ακόμα και θα πρέπει να δούμε τι αποφάνθηκε τελικά και το Συμβούλιο για τους συμβιβασμούς που πετύχαμε στην τρομερή διάλογο, αλλά ε, Γενικώ πώ σημειώνεται πρόοδο, από ό,τι φαίνεται. Ένα άλλο άρθρο τώρα. Όπου ζητούμε την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε ό,τι αφορά το άρθρο που προτείνεται για την Ευρωπαϊκό Ένταλμα Έρευνας και σχετική νομική αρρωγή σε ό,τι αφορά λοιπόν ε, διάφορα στοιχεία όπως για παράδειγμα η, η ανακατασκευή της ε, του ζημιού του που διεξήχθη το έγκλημα κτλ. Εκεί λοιπόν... Ε, ε από εδώ λοιπόν ε, εξαρτώμαστε πολύ από την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με το τι είναι νομικά απαραίτητο μετά την πρόσβαση στο δικηγόρο που ασφαλώς ε, αυτό είναι καθοδηγητικό στοιχείο σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή. Φαίνεται λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει αυτή η σειρά Ενδεχομένως να υπάρχει όμως ένα νομικό κενό, αν δεν αναφερθούμε ρητά σε καταστάσεις όπου τρίτες χώρες ζητούν τέτοια μέτρα ή αν εμπλέκεται μια χώρα στην οποία ισχύουν τέτοιες προδιαγραφές. Θα περιμένουμε λοιπόν και το πόρισμα της νομικής ανάλυσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να συνεχίσουμε και σε αυτό το άρθρο. Και νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό Έχουμε επεξεργαστεί σχεδόν όλα όσα σκοπεύαμε να επεξεργαστούμε κατά την Ολλανδική Προεδρία και 3 Μαΐου προβλέπεται ο επόμενος τριμερής διάλογος. Ε, αυτό για να ε, αναφερθούμε και σε μια άλλη πρωτοβουλία που είχαμε λάβει πέρσι σε ό,τι αφορά μια μερικά δικτύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το ποιε θα είναι οι συνέπειε των τροπολογιών που προτείναμε σε σύγκριση και με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε λοιπόν τη μελέτη αντικτύπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν υπήρχε όμω σχετική ανάλυση μελέτη αντικτύπου για τις συνέπειε των σημαντικών τροπολογιών μας. Ε, έτσι θα εστιαστούμε όχι μόνο στο οικονομικό κόστος, αλλά και στις συνέπειες ε, των τροπολογιών μας για τα θεμελιώδη δικαιώματα και κυρίως για τα κοινωνικά δικαιώματα. Άρα θα υπάρχει μια ισορροπημένη μελέτη αντικτύπου και αυτό που είναι σημαντικό για μας είναι να υπάρχει περαιτέρω διάλογος με το Συμβούλιο όταν θα είναι έτοιμο το κείμενο, για να ξέρουμε τι συζητάμε. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό αναμένουμε ένα πρώτο σχέδιο, όχι το τελικό σχέδιο, ένα πρώτο σχέδιο να το έχουμε στη διαθέσή μας ε, μέσα Απριλίου στα μέσα Απριλίου για την μέθοδη τύπου και μια στρατηγική συνάντηση των σκιωδών για να συζητήσουμε τι θα κάνουμε, πώς θα συνεχίσουμε. 9 Απριλίου, αρκετά πριν λοιπόν, την τον επόμενο τριμερή διάλογο. Θα παρουσιάσω στους σκιώδες λοιπόν στην χρονική στιγμή αυτή. Η γραμματεία θα παρουσιάσει τη μέθοδη αλλά εγώ θα προσπαθήσω να καταρτήσω ένα έγγραφο εργασίας που θα περιλαμβάνει όλες τις εναλλακτικές και μετά θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε με ανοιχτό πνεύμα, όπως έχουμε κάνει και ως τώρα άλλωστε, και ελπίζω να συνεχίσουμε με την ίδια ομόνια και ομοφωνία, όπως έως τώρα. Σε ό,τι αφορά τώρα το ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί την επόμενο ήμιση της Ολλανδικής Προεδρίας, επειδή σημειώνεται πρόοδος, μία λύση θα ήταν να βρεθούν λύσεις για όλο το πακέτο μέσα στην Ολλανδική Προεδρία. Είναι αρκετά φιλόδοξο σχέδιο, αλλά γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι τόσο σημαντική η συνάντηση στις 9 Απριλίου και πραγματικά ελπίζω να παρευρεθούν και να συμμετάσχουν οι συνάδελφοι. Γιατί αν δεν ε, συμμετάσχουμε όλοι, πώς θα αποφασίσουμε τι θα κάνουμε στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Ντένις. Και εγώ ελπίζω να είναι όλοι και όλες παρούσεις παρόντες. Να δώσω τώρα το λόγο σε όλους τους κοιόδους που είναι εδώ. Ε, και η μόνη που είναι εδώ είναι η κυρία Ζίπελ, η υποφαινομένη δηλαδή, σκιώδηση συγγήτρια από την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, η οποία θα μιλήσει και στα γερμανικά σήμερα. Να ευχαριστήσω καταρχάς τον Τένις για τη δουλειά του. Να σας ευχαριστήσω και τους υπόλοιπους σκιώδες συζητητές, γιατί ως τώρα πραγματικά ήταν εξαιρετική και επικοδομητικότητα συνεργασία. Όπως ανέφερε και ο Ντένις στα εισαγωγικά του σχόλια, σε κάποια σημεία έχουμε πετύχει μια προσωρινή τουλάχιστον συμφωνία που είναι πάρα πολύ σημαντική για μας ως Κοινοβούλιο. Σε σύγκριση με το σχέδιο οδηγίας έχουμε προσθέσει ένα νέο άρθρο για τις αρμόδιες αρχές σε ό,τι αφορά την, το αίτημα συμμετοχής στα έξοδα τα δικαστικά. Και θεωρούμε ότι η αυτή η απόφαση θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τον υπολογισμό τεχνικών και διαδικαστικών εξόδων και σε ό,τι αφορά τα έξοδα για την αποτελεσματικότητα της εκδίκασης θα πρέπει να συνυπολογιστούν και ότι αυτό δεν θα αλλάξει ως ε, διαπραγματευτική θέση. Θα υπάρξει και ένα περαιτέρω άρθρο για την επέκταση της νομικής αρρωγής. Όλα αυτά, και το υπάλληλο άλλωστε και ο Ντένις, όλα αυτά είναι προσωρινά ωστόσο. Αυτό που εκκρεμεί ακόμα είναι η συμφωνία, η συνένεση των εθνικών κυβερνήσεων. Άρα δεν είμαι καθόλου βέβαιη κατά πόσον θα συνεχίσουν να υφίστανται μετά τη συζήτηση με τα κράτη-μέλη, γιατί ποτέ κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρο ή ενδεχομένως αν θα αποδυναμωθούν, θα απορριφθούν 100%. Ελπίζω και στο σημείο αυτό όμως να υπάρχει μια επικοδομητική διάθεση και να προχωρήσουμε έτσι επικοδομητικά. Πέρα από τις προσωρινές αυτές συμφωνίε. συμφωνίες υπάρχουν και κάποια άλλα εκκρεμή στοιχεία, τα οποία ήδη τα έδειξε ο συνάδελφος Ντένις για τα γενικά δικαστικά έξοδα και την αρρωγή ως προς αυτά και όπως όλοι οι σκιώδεις, ε, φαντάζομαι είμαι και εγώ α, περίεργη να δω ποια θα είναι τα αποτελέσματα της μελέτη αντικτύπου. Μπορεί να ενισχύσουν τη θέση μας. Ε, γι' αυτό λοιπόν προσβλέπω στην περαιτέρω μελλοντική επικοδομητική συνεργασία με τον Τένις και τους άλλους ε, εισηγητές και σε μια καλή συνεργασία και με το Συμβούλιο. Σας ευχαριστούμε κυρία Σίπελ, λέει η Πρόεδρος. Τώρα, Μήπως θα ήθελε και κάποιο άλλο θεσμικό όργανο να πάρει το λόγο για να μιλήσει το θέμα αυτό. Δεν υποχρεούστε ασφαλώς μόνο εφόσον το επιθυμείτε. Αν θα ήθελε το Συμβούλιο, έχει το λόγο. Uh, ναι, θα μπορούσα να πω δύο λόγια. Αλλά νομίζω θα πω τα ίδια με τον εισηγητή περίπου. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν κυρία Πρόεδρε. Δεν νομίζω ότι είναι γνωστό ότι η γενική ε, προσέγγιση Συμβουλίου διαφέρει από αυτήν του Κοινοβουλίου. Εμείς ε, περιοριζόμαστε ε, στο πεδίο εφαρμογής αυτή τη οδηγία, εσεί θέλετε να επεκτείνετε και στην έκτακτη νομική συνδρομή για τα άτομα στα οποία δεν παρέχονται εγγύηση. Ωστόσο, η Προεδρία μαζί με τον εισηγητή και του κοιόδες καταβάλει προσπάθειες για την εξέβρεση πρακτικών λύσεων ώστε να βρούμε ένα κείμενο που θα ήταν αποδεκτό για του δύο συνομοθέτες και να μην συζητάμε επί τη αρχή, όπω είπε και ο κύριο Ντε έχουν, γίνει μέχρι τώρα δύο τριμερεί διάλογοι. Θεωρούμε ότι ήταν πολύ επικοδομητικό το κλίμα και υπήρξε σαφής προθυμία γεφύρωσης του χάσματος και να γίνουν συμβιβασμοί και από τις δύο πλευρές. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ντεγιόν και τους κοιότητες ε, εισηγητές γιατί ήταν πολύ επικοδομητική η στάση τους ε, στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Σε αυτή τη φάση είναι δύσκολο να προβλέψουμε τι θα συμβεί τους ε, προσεχείς μήνες και νομίζω δεν χρειάζεται καν να σας πω ότι πολλά θα εξαρτηθούν από την έκβαση της μελέτης αντικτύπου που διεξάγει το Κοινοβούλιο του παρόντος, στρατηγικά συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και βέβαια και από τις απόψεις των κρατών μελών. Η Προεδρία θα κάνει κάθε προσπάθεια ώστε να προχωρήσουν πραγματεύσει το πολύ σημαντικό αυτό ζήτημα. Προσβλέπουμε και στην μελλοντική συνεργασία μας. Ευχαριστώ. Thank you very much for these few words from the council. Ακούσαμε λοιπόν λίγα λόγια και από το Συμβούλιο. Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα φαίνεται να μην θέλει το λόγο. Άρα μπορούμε να ολοκληρώσουμε το σημείο αυτό και να περάσουμε ευθύ αμέσω στο σημείο 5 της μερισιάς διάταξης, παρουσίαση από τον Ιωάννη Δημητρακόπουλο, της έκθεσης ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σε επαγγελματικό επίπεδο προκλήσεις για την επίτευξη ισότητας ε, για τους ε, ΛΟΑΔ. Χαιρόμαστε πολύ που είστε εδώ και βέβαια περιμένουμε να ακούσουμε πολύ ενδιαφέρον την παρουσίασή σας. Παρακαλώ το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, καταρχά να ευχαριστήσω για την πρόσκληση εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για να σα παρουσιάσουμε το έργο μα σε σχέση με την κατάσταση των ε, ε, λεσβιών, ομοφυλοφίλων, διεμφυλικών, ε, φιλομεταβατικών και λοιπόν συντομία ΛΟΑΔ. Σίγουρα μπορεί να διαφορετική σεξουαλική ταυτότητα αυτών των ατόμων, όμω έχουν τα ίδια δικαιώματα και πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα. Έχουν το ίδιο δικαίωμα να ζουν ε, με αξιοπρέπεια, να μην φοβούνται και να μην υφίστανται διακρίσει. Ε, μέχρι τώρα η δουλειά που έχουμε κάνει δείχνει ότι παρά τη σημαντική πρόοδο ε, στην νομοθεσία, στην πολιτική, πολλά ακόμη πρέπει να γίνουν για να πετύχουμε. Ε, αυτή την ισότητα επιτόπου. Έχουμε ξεκινήσει να συλλέγουμε ενδείξεις ε, σε, ό,τι αφορά ε, την κατάσταση των ΛΟΑΤ. Ξεκινήσαμε 9 χρόνια πριν, μόλις θεσπίστηκε ο οργανισμός μας και αυτό ήταν κατόπιν συγκεκριμένου τίματος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καταρχάς εξετάσαμε και κάναμε και μια συγκριτική ανάλυση που δημοσιεύτηκε ήδη το 2010, τους νόμους και πολιτικές που επηρεάζουν ε, τις ζωές ε, των ε, ατόμων ΛΟΑΔ. Πιο πρόσφατη επικαιροποίηση είναι αυτή του Δεκεμβρίου 2015, η τρίτη επικαιροποίηση που δείχνει τις τάσεις, αναφέρει τις βελτιώσεις, αλλά επισημαίνει και τα κενά και τις αδυναμίες. Αυτή τη στιγμή περιλάβαμε συγκριτική ανάλυση των δικαιωμάτων και των των ατόμων ε, intersex που τους είχαμε ε, μέχρι στιγμής ε, κατά κάποιο τρόπο παραμελήσει. Το 2013 επίσης δημοσιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα της ευρύτερης μέχρι στιγμής έρευνα. Πάνω από 93.000 ε, άνθρωποι ε, ε, από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασαν τις ανησυχίες τους, μας έδωσαν τις προσδοκίες τους και την προηγούμενη εβδομάδα παρουσιάσαμε τα πορίσματα της τελευταίας μας έρευνας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό είναι και τελευταίο, αν θέλετε, κομμάτι του παζλ και επιβιώνει και τις, ε, τα πορίσματα της έρευνας που έδωσε, είπαμε, ε, φωνή σε, όπως είπα, πάνω από 93.000 ανθρώπους από όλο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ όμως αυτό που θέλω τώρα να σας πω δίνει ουσιαστικά φωνή σε αυτούς που έχουν πλέον ε, το καθήκον στην άλλη πλευρά ε, να φέρουν σε πέρας πολιτικές. Πάνω από χίλιοι δημόσιοι υπάλληλοι, γιατροί, ε, εκπαιδευτικοί, αστυνομικοί, ομάδες επαγγελματιών οι οποίοι γνωρίζουν από πρώτο χέρι και καλύτερα από άλλους την κατάσταση. Πρώτα απ' όλα να δούμε ποιοι είναι οι φραγμοί, ποια είναι τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι λάβημα και στον τομέα τη εκπαίδευση, τη υγειονομική περίθαλψη και τη επιβολή ε, του νόμου. Δεύτερον, επίση θέλουμε να δούμε τι ε, άποψη έχουν οι ίδιοι των κλάδων αυτών και πώ μπορούν να προωθήσουν ε, τα δικαιώματα των ΛΟΑΔ. Με εστιάσαμε σε τομεί όπου μέχρι στιγμή η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία δεν παρέχει προστασία από τη διακρατική μεταρρύθμιση λόγω γεννητή προσανατολισμού. Θέλαμε να δούμε αν τα αποτελέσματα τη έρευνά μα που έδειξαν ότι οι άνθρωποι ΛΟΑΔΜΑ βιώνουν παρενόχληση και διακριτική μεταχείριση όχι μόνο στην εκπαίδευση ή στον χώρο τη εργασία του, αλλά και σε άλλου πολύ σημαντικού τομεί τη κοινωνική ζωή, αν αυτά τα αστεία μπορούμε να τα επιβεβαιώσουμε. Και πράγματι, με τα πορίσματά μα βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλήματα στην εκπαίδευση, στην υγεία, και σε σχέση με την αστυνομία για τους ΛΟΑΔΜΑ και ε, επίσης ε, είδαμε ότι χρειάζεται ανάγκη να ε, υπάρχει μια οδηγία, ε, οριζόντια οδηγία για την ισότητα μεταχείριση. Να ξεκινήσω με τις απαντήσεις των δημόσιων υπαλλήλων αξιωματούχων που είναι υπεύθυνοι για τη χάραξη και εφαρμογή των πολιτικών ισότητας. Οι συνεντεύξεις έδειξαν ότι περισσότεροι είναι προσιλωμένοι στην βελτίωση της κατάστασης των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ, υπεγράμμισαν ότι θεωρούν ε, την νομοθεσία και πολιτικέ περισσότερε τη Ένωση σε σημαντικό κινητήριο μοχλό αλλαγής στις χώρες τους ε, άρα επηρεάζει η ευρωπαϊκή πολιτική το εθνικό επίπεδο, θεωρούν επίσης χρήσιμες αυτές τις ε, πολιτικές και στην καθημερινή τους δουλειά. Πιστεύουν ότι είναι θετική δράση τη Ένωση, ωστόσο τονίζουν ταυτόχρονα τη, σημαντική, τη, σημασία δύο άλλων πολύ σπουδών παραγόντων που είναι η δημόσια υποστήριξη από τους πολιτικούς ηγέτες και η ισορροπημένη κάλυψη από τα ΜΜΕ, δύο στις χώρες όπου είναι ακόμη αμφισβητούμενο το θέμα της ε, ταυτότητας των ΛΟΑΔΜΑ. Υπάρχουν επίσης προκλήσεις που επιμένουν. Και υπάρχουν δύο ε, εμπόδια πολύ σημαντικά. Πρώτα απ' όλα, εμέν προκαταλήψεις και η έλλειψη ανεκτικότητας, ιδίως στα νότια και δυτικά κράτη της Ένωσης. Και επίσης ε, βλέπουμε ότι σε όλα τα κράτη-μέλη ε, υπάρχουν και προκαταλήψεις. Οι δημόσιες αρχές δεν επενδύουν σε πολιτικές ισότητας εάν οι δικαιούχοι δεν είναι ορατοί, δεν φαίνονται ή δεν μιλάνε και δεν διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Έρχομαι τώρα στην εκπαίδευση. Ε, ήρθαμε συνεντεύξεις με ε, γυμνασιάρχες, λυκιάρχες ε, και εκπαιδευτικούς που μας μίλησαν ότι υπάρχει ε, εκφοβισμός, υπάρχουν κάποια μέτρα γενικά και κατά το εκφοβισμού που όμως δεν αντιμετωπίζουν τις πιο ειδικέ μορφές, δηλαδή όταν μιλάμε συγκεκριμένα για φοιτητές ΛΟΑΔΜ. Ένας δάσκαλος όμως είπε και νομίζω ότι αυτό αντικατοπτρίζει από όλων άλλων η βία στα σχολεία και παραπέμπω δεν είναι το σημαντικότερο πρόβλημα. Αυτό που είναι σημαντικότερο σήμερα είναι ένα ομοφοβικό κλίμα με επαναλαμβανόμενες ε, ε, προσβολές που θεωρούνται κάτι τετριμένο και καθημερινό, που όμως ε, δημιουργούν μεγάλο άγχος για τους ε, φοιτητές ΛΟΑΔ. Πολλοί εκπαιδευτικοί μίλησαν και για την έλλειψη εκπαιδευτικού υλικού, για το σεξουαλικό προσανατολισμό και την γεννήσια ταυτότητα ή για την ισότητα των ατόμων ΛΟΑΔ. Δεν είναι στη διδακτέα ηλίτσα, όχι στο πολίτη. Επίσης παραπονέθηκαν ότι δεν υπάρχει επαρκή εκπαίδευση, ούτε επαρκή εργαλεία για τη στήριξη των φοιτητών ΛΟΑΔ που αντιμετωπίζουν προβλήματα μαθήματα στο σχολείο. Τα κράτη-μέλη ναι μεν έχουν ε, εφαρμόσει και σχεδιάσει μέτρα κατά το εκφοβισμό ώστε να υπάρχει ένα πιο υποστηριστικό κλίμα για ΛΟΑΔΜΑ, μαθητές αλλά και εκπαιδευτικούς ε, στην Κύπρο, στην Ελλαδία, στον Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες χώρες. Πρέπει να γίνουν πολλά όμως ακόμη, ώστε να μπορούν οι ήδη εκπαιδευτικοί να στηρίξουν τους ε, σπουδαστές ΛΟΑΔΜΑ και κοινωνικά στα σχολεία. Περνάω τώρα στην υγειονομική Πέριθλο, στον τομέα τη υγεία. Πολύ λεπτό τομέα. Ε, απαιτείται επαγρύπνηση ώστε όλοι να αντιμετωπίζονται ε, με τον ίδιο τρόπο και να έχουν το στο δυνατό επίπεδο ε, περίθαλψη οι ΛΟΑΔΜ πρέπει να αντιμετωπίζονται ω ασθενεί με την ίδια προσοχή, με τον ίδιο σεβασμό όπω όλοι. Σε κάποιε χώρε πάντα, όπω Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ιταλία, ε, Λετωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Πολωνία, με έκπληξη ακούσαμε από κάποιου από του γιατρού με του οποίου είχαμε συνέντευξη επιχειρήματα ε, που δείχνουν ότι κάποιοι από του συναδέλφου του θεωρούν νόσο ε, την ομοφιλοφιλία. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα για το πώς θα αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους γιατροί ασθενείς, οι οποίοι το λένε κιόλας. Επίσης, πολλοί από τους γιατρούς ε, είπαν ότι δεν υπάρχουν ειδικέ πολιτικές, μέσα, εκπαίδευση για την καλύτερη υποστήριξη των ΛΑΜ, ιδίως στα κέντρα και στα νοσοκομεία. Όταν Βλέπουμε τώρα τα ε, δημοφιλικά ζητήματα. Υπάρχουν γιατροί οι οποίοι δικεύονται σε αυτόν τον τομέα και είπαν ότι δεν υπάρχουν εξειδικευμένε ιατρικέ υπηρεσίε ούτε και ευαισθητοποίηση και συνειδητοποίηση των γιατρών για τι συγκεκριμένε προκλήσει ε, των ε, ανθρώπων αυτών. Χειρουργική για τον προσδιορισμό του φύλου είναι προβληματική σε πολλά κράτη-μέλη. Στη Λιθουανία, για παράδειγμα, Μόνο στο εξωτερικό μπορούν να ε, χειρουργηθούν οι άνθρωποι αυτοί. Και έπειτα πρέπει να γίνουν δίκες για να μπορέσουν να αλλάξουν και τα ε, έγγραφα, τα προσωπικά τους, ταυτότητες και Τα λοιπά. Τώρα, επιβολή νομοθεσία δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Σε πολλές χώρες είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούν αστυνομικοί οι οποίοι ε, θα ήθελαν να δώσουν συνέντευξη για θέματα που αφορούν τους climate. Αυτό δείχνει πιστεύω το κλίμα που επικρατεί. Όσοι απάντησαν πάντως είπαν ότι δεν υπάρχει παρκή ευστοποίηση στην ε, βαλωτότητα των ατόμων αυτών ε, που υφίστανται και ε, είναι θύματα εγκλημάτων μίσους. Είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μας ότι η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι πιο Καλή έχουμε μία οδηγία του 2012 που λέει ότι πρέπει να εκτιμηθούν καλύτερα οι ανάγκες, να λαμβάνονται υπόψη τα προσωπικά χαρακτηριστικά του θύματος και το είδος του εγκλήματος. Αυτό μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ ε, θύματα εξώπινων πράξεων που είναι ΛΟΑΔΜΑ. Βέβαια, Κάποιοι εξωματούχοι με τους οποίους ε, ήρθαμε σε επαφή δεν αναγνώρισαν ή υποτίμησαν την κλίμακα και το είδος ε, αυτών των συμβάντων ε, και των πράξεων βίας ή μίσους κατά τον ΛΟΑΔΜΑ. Στις περισσότερες χώρες οι αστυνομικοί μίλησαν για έλλειψη συστηματικής και αποτελεσματικής εκπαίδευσης των αρχών για να αντιμετωπίσουν αυτά τα εγκλήματα, τι εξώπαινε αυτέ τι πράξει, γιατί δεν υπάρχει ε, ενδιαφέρον, η καλή θέληση, υπάρχουν περιορισμένοι πόροι, αλλά σε κάποια κράτη-μέλη όπω Αυστρία, Κροατία, Δανία, Λανδία, Ολλανδία, Ενωμένο Βασίλειο, αστυνομικοί είπαν ότι λαμβάνονται σημαντικέ πρωτοβουλίε από την απλή αύξηση τη ευαισθητοποίηση μέχρι εξειδικευμένη παροχή εκπαίδευση και συνεργασία μεταξύ αστυνομικών αρχών και κοινωνία των πολιτών και συγκεκριμένων οργανώσεων λάδου, Για τη βελτίωση τη αναφορά ε, τέτοιων αξιόπινων πράξεων και για τη βελτίωση τη ασφάλεια των λάδων. Ολοκληρώνοντα, θα ήθελα να ε, διαλώσω ότι στηρίζουμε δράση για την πρόθεση της ισότητας. Λοιπόν, είχαμε μια σχετική δημοσίευση πέρυσι ε, από την Κομισιόν, ένα κατάλογο που δεν είναι ακριβώ ο δικό χάρτη πιεστή στο Κοινοβούλιο, πάντω είναι ένα σημαντικό ε, πακέτο μέτρων και θα πρέπει να το θεωρήσουμε ένα σταθμό. Τελευταία έκθεση του οργανισμού μα ε, που διατίθεται στην αίθουσα περιλαμβάνει κάποιε απόψει και απευθύνεται στα κρατμέλη. Πιστεύω ότι μπορείτε να βρείτε χρήσιμα τα όσα αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο και ολοκληρώνοντα να αναφέρω τρει από τι απόψει αυτέ που θεωρώ πολύ σημαντικέ. Πρώτον, πρέπει να ενθαρρύνουμε την προβολή των ΛΟΑΤ. Πολιτική οικονομική στήριξη, παραδείγματο χάρη, για τι παρελάσει Pride κτλ. Δεύτερον, να δώσουμε το καλό παράδειγμα. Ε, με ελέγχου ε, καλή ε, ισότητα, μάλλον και με τι διάφορε στρατηγικέ ή κώδικε καλή συμπεριφορά, με μετρήσιμα αποτελέσματα. Και τρίτον, να ετοιμαστούμε για το μέλλον, να προετοιμάσουμε τους εκπαιδευτικούς, να τους δώσουμε μέσα, ε, δεξιότητες για να μπορούν τα σχολεία τους να τα μετατρέψουν σε ένα πιστορικτικό περιβάλλον, ώστε όλα τα παιδιά και το, το, τα παιδιά ΛΟΑΔΜΑ να τα προετοιμάσουν να ζουν σε μια κοινωνία ε, όπου γίνεται σεβαστή η, αξιο, η αξιοπρέπεια, το κάτω δικαίωμα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και βέβαια τα δικαιώματα ανθρώπων που ανήκουν σε μειονότητες. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, Ευχαριστώ πολύ κύριε Δημήτρα Κόπουλε. Θεωρώ ότι πρόκειται για πολύ σημαντική έκθεση, διότι αν δούμε γύρω μας, ορισμένες φορές νιώθουμε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, διότι υπάρχουν πολιτικοί, ηθοποιοί και άλλοι διάσημοι, οι οποίοι δηλώνουν δημοσίως την ομοφιλοφιλία τους και λέμε ότι αν είναι δυνατόν κάτι τέτοιο, προφανώς δεν υπάρχουν προβλήματα. Γνωρίζουμε όμως από άλλες εμπειρίες ότι υπάρχουν προβλήματα και η έκθεσή σας σαφώς καταδεικνύει που έγκυται αυτά τα προβλήματα στους διάφορους τομείς. Επομένως, πρόκειται για ε, εργασία η οποία είναι πολύ χρήσιμη για να μπορέσουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να ξεπεράσουμε τις ανισότητες που αντιμετωπίζουν οι ΛΟΑΔ στην κοινωνία μας. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος συνάδελφος θέλει να λάβει το λόγο ή Τζιν Λάμπερτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Και θα ήθελα να μου πείτε λίγα περισσότερα για την ε, ε, άποψή σας ε, Πού νομίζω ότι βρίσκεται το παιχνίδι μεταξύ ε, της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας η οποία ε, σημαίνει και ευθύνε για τους εργοδότες ε, και για φορείς ποιότητες οι οποίοι πρέπει να διασφαλίσουν ότι εμφαρμόζεται αυτή η νομοθεσία. Και έχουμε επίσης και ε, δυνατότητες χρηματοδότησης που μπορούν να βοηθήσουν στους ανθρώπους στον χώρο της εργασίας να αντιμετωπίσουν τη διαφορετικότητα και μάλιστα σωστά. Πώς μπορείτε λοιπόν να θεωρείτε ότι θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε περισσότερο αυτό για να αλλάξουμε την οτροπία της κοινωνίας. Διότι αν αναφερόμαστε σε νοοτροπία των αστυνομικών δυνάμεων, στην παιδεία, στη δημόσια διοίκηση και στην ε, περίθαλψη, υπάρχει νομοθεσία που ισχύει για αυτούς στον χώρο της εργασίας. Πώς μπορούμε λοιπόν να ε, το περάσουμε αυτό από το χώρο της εργοσίας ευρύτερα στην κοινωνία, χρησιμοποιώντας το ως βάση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιουρέκ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας θέσω αρκετές ερωτήσεις. Αυτή η μεσοφελική προσέγγιση. Ε, την κατηγορία αυτή την παραλείψατε στην παρουσίασή σας σκοπίμως ε, ή η κατηγορία αυτή είναι μια κατηγορία που δεν είναι αρκετά γνωστή. Και κάτι ακόμα το οποίο θα ήθελα να θίξω. Η άποψή σας για τα δημοψηφίσματα στη Σλοβακία και στη Σλοβενία. τα οποία αφορούσαν αίτημα τη κοινότητα στο ΛΟΑΔΜ για τα σχολεία, παραδείγματι. Το δικαίωμα στην εργασία είναι καθολικό δικαίωμα. Αλλά η περιγραφή της πραγματικότητας που μας κάνατε με ανησυχεί λίγο, διότι φαίνεται να αποστασιοποιούμαστε από τις χριστιανικές αρχές η οποία είναι και, ε, οι οποίες είναι και εγγεγραμμένες στη συνθήκη. Και υπάρχει μια αρνητική προσέγγιση ε, στις πράξεις των ομοφιλοφίλων, όχι στην τάση για ομοφιλοφιλία. Μπορεί να έχουμε μια κοινότητα της οποίας τα μέλη προσπαθούν να απέχουν από οποιαδήποτε σεξουαλική δραστηριότητα και θέλουν απλώς να παραμείνουν ε, αγνοί. Ποια είναι η άποψή σας ε, για αυτή την προσέγγιση στη ζωή. Και αυτό είναι μια μορφή εκδήλωσης σεξουαλικότητας μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να βελτιώσουν την ηθική τους γιατί ε, ζουν σε κοινότητες οι οποίες δεν προωθούν οποιαδήποτε συγκεκριμένη ε, προσέγγιση. Αυτά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να κάνω κάποιες συμπληρωματικές ερωτήσεις από δική μου πλευρά. Όταν μιλάμε για τους ΛΟΑΔΜΑ ή τους ΛΟΑΔΑ, Αναφέρατε το σημείο της ιατρικής παρακολούθησης και περιθαλψής, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους μεσοφιλικούς και τους διαφιλικούς. Θα ήθελα να ξέρω πού πιστεύετε ότι υπάρχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα με τους γιατρούς. Είναι πιο πολύ ο σωματικός ε, παράγοντας ή πιο πολύ η ψυχολογική συνέπεια. Και τι στοιχεία λαμβάνονται υπόψη τι συμβουλές δίδονται και πολύ δύσκολο βρίσκω το θέμα που θίξατε σε σχέση με την ανατροφή. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρόκειται να έχουμε ίσα δικαιώματα για όλους τους ανθρώπους και ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και οι μειονότητες έχουν ίδια δικαιώματα όπως οι υπόλοιποι πολίτες. Αλλά θα συνεχίσει αυτό να αποτελεί πρόβλημα όσο στα στις σχολικές ε, ή και στα σπίτια μας ε, α, λέμε ότι κάποιος είναι ομοφιλόφιλος και το λέμε σαν βρισιά. Χωρίς να ξέρει το άτομο που χρησιμοποιεί τη λέξη αυτή, τι κρύβεται πίσω από τη λέξη αυτή. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να μας πείτε αν έχετε κάποια σύσταση, κάποια πρόταση σε ό,τι αφορά το εκπαιδευτικό υλικό, σε ό,τι αφορά τα... τη σχολική ύλη και μάλιστα σε όλα τα μαθήματα, σε ό,τι αφορά τα εγκλήματα με βάση τα εγκλήματα μίσους, θα ήθελα να αναφερθώ στις ε, στατιστικές σε ό,τι αφορά την εγκληματικότητα. Ξέρουμε ότι σε κάποια κράτη δεν υπάρχουν πραγματικά στατιστικά στοιχεία ε, που να καλύπτουν τις ακροδεξιές εκφάνσεις του εγκλήματος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και πιστεύετε ότι υπάρχουν τουλάχιστον σε κάποιες χώρες τέτοια στοιχεία σε ό,τι αφορά τα εγκλήματα ως ακραία ένδειξη απόρριψη των ΛΟΑΔ ή πιστεύετε ότι δεν καλύπτονται στα στατιστικά στοιχεία τα εγκλήματα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να πω καταρχάς να ξεκινήσω αναφερόμενο σε κάποια από τα σημεία τα οποία ήδη ανέφερα ελπίζω αρκετά σαφώς στην παρουσίασή μας σε ό,τι αφορά το αίτημα για μία οριζόντια, μάλλον μία οδηγία αποτελεσματική για την οριζόντια αυτή διάσταση. Οι 43 και 48 οδηγίες, όπως σας είπα, έχουν θέσει μια ιεραρχία. Έχουν θέσει την φίλη και την εθνοτική προέλευση που προστατεύονται πολύ καλύτερα από όλα τα κοινωνικά ζητήματα, από την αναπηρία, την ηλικία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό που δεν καλύπτονται, δεν προστατεύονται εξίσου. Η πρόταση που έγινε το 2008 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρούμε ότι εν μέρη θα κάλυπτε αυτό το φάσμα που υπάρχει τώρα. Η νομοθεσία δεν έχει να κάνει μόνο με την πρόληψη και την επιβολή ποινών έχει να κάνει και με την ευαισθητοποίηση, την εκπαίδευση για την... ένα υπόδειγμα για το τι θα πρέπει να κάνουμε στην καθημερινή μας ζωή. Και θα μπορούσε να αποτελεί λοιπόν ένα σαφέ μήνυμα από πλευρά των θεσμικών οργάνων τη Ευρωπαϊκή Ένωση η έγκριση μια τέτοια οδηγία, την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί μάλλον το ότι θα πρέπει όλα τα στοιχεία να προστατεύονται ε, εξίσου σε ό,τι αφορά την ε, ίση μεταχείριση. Έχουμε λοιπόν κάποιες πολύ σημαντικούς τομείς για όλους που καλύπτουν την καθημερινή μας ζωή, ιδιαίτερα για τους ε, νεότερους. Και θα ήταν περίεργο η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην κάνει κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια αναγνωρίζοντας φυσικά ότι η πρωτεύουσα αρμοδιότητα είναι στα χέρια των κρατών μελών για τέτοια ζητήματα. Αλλά θα ήταν λίγο παράλογο να μην σπρώξει τα κράτη-μέλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προστατεύσει καλύτερα τα άτομα που ανήκουν σε μειονότητες, προκειμένου να τη χάνουν ίσες μεταχειρήσεις. Δεν ξέρω κατά πόσον αναφέρθηκα σε δημοψηφίσματα στα κράτη-μέλη, αλλά φυσικά και τα κράτη-μέλη έχουν δικαίωμα να διοργανώσουν δημοψηφίσματα με όποιο τρόπο το επιθυμούν για να πραγματευτούν διάφορα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικογενειακή πολιτική όσο εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Δημοθεσίας και των Ευρωπαϊκών Συνθήκων. Αναγνωρίζω δε ότι το θέμα των μεσοφιλικών το δεν το έχουμε πραγματευτεί στο παρελθόν και γι' αυτό λοιπόν η μελέτη που παρουσίασα σήμερα η οποία ε, ολοκληρώθηκε πριν από 1,5 χρόνο σε ό,τι αφορά τη συλλογή των στοιχείων, δεν τους περιλάμβανε τους μεσοφιλικούς. Ξεκινήσαμε τη συλλογή στοιχείων φέτος και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση με πιο μεγάλο επίπεδο λεπτομέρειας για τα εγκλήματα μίσους και τα στατιστικά στοιχεία. Προτού εξετάσουμε το κατά πόσον τα εγκλήματα μίσους κατά τον ΛΟΑΔ καλύπτονται από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, θα πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να εξετάσουμε κατά πόσο η επιβολή του νόμου έχει τα απαραίτητα εργαλεία για να καταγράψει τέτοιου είδου εγκλήματα. Μίλησατε για τη Γερμανία, τη Γαλλία, όπου τουλάχιστον κατά από το παρελθόν τα εγκλήματα μίσους καταγράφονται μόνο εφόσον ήταν ε, και προέρχονταν από εξτρεμιστικές ακροδεξίες οργανώσεις και τάσεις. Είναι σημαντικό φυσικά αυτό, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς ε, καταγράφει η αστυνομία κάθε κράτος μέλους τα εγκλήματα μίσους. Ε. υπάρχει, για παράδειγμα, σχετικό πίνακα για να αναφέρονται και τα αίτια του εγκλήματος μίσους και τα διάφορα είδη δραστών. Υπάρχουν διάφορα στάδια, θεωρούμε. Είναι το θέμα της ε, αναφοράς του εγκλήματος μίσους, γιατί οι πιο, πολλοί, οι πιο πολλές μειονότητες, οι ΛΟΑΔ, ακόμα και οι γυναίκες που δεν είναι η μειονότητα, ακόμα λοιπόν και οι γυναίκες θεωρούν ότι είναι δύσκολο να απευθυνθούν στις αρχές επιβολής του νόμου και να αναφέρουν το έγκλημα. Άρα είναι σημαντικό να υπάρχει πραγματικά αναφορά. Το πρώτο βήμα είναι αυτό. Όταν λοιπόν γίνεται η αναφορά, οι αστυνομικέ δυνάμει θα πρέπει να είναι έτοιμε, και να έχουν τα σωστά, τους σωστές πίνακες για να μπορούν να καταγράψουν σωστά α, το έγκλημα. Και φυσικά τρίτο βήμα είναι η δίωξη. Θα πρέπει όλα αυτά όμως να είναι συντονισμένα και θα συνεργαστούμε με την επιβολή του νόμου, με τις δικαστικές αρχές για να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την αφορά την καταχώρηση των εγκλημάτων μίσους προκειμένου να περιλαμβάνεται και η φύση του εγκλήματος ακριβώς. Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Κατά τη συζήτηση σε διάφορες περιστάσεις ε, αναφέρθηκε η οδηγία ίσης μεταχείρισης. Δεν είναι άλλο μυστικό ότι εδώ στο Κοινοβούλιο πολλοί κόσμος ε, τη χρησιμοποιεί την οδηγία για να τονίσει ότι ο κάθε πολίτης ε, στην Ένωση έχει τα ίδια δικαιώματα. Ακόμα και η Επιτροπή που παρουσιάσει την πρόταση εκείνη είναι υπέρ των σημείων αυτών. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη αυτά τα στοιχεία που αναφέρθηκαν σήμερα το απόγευμα στη συζήτηση, να στραφούμε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ρωτήσουμε κατά πόσον θα ήθελε να μας δώσει κάποιες ιδέες σε ό,τι αφορά την ίση μεταχείριση. Χαίρετε. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για την έκθεση αυτή και την Επιτροπή ΛΥΠΕ που την έβαλε στην ημερήσια διάταξη. Όσον αφορά την οδηγία αυτή, θα γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιέζει πάρα πολύ για τα ίσα δικαιώματα και αυτό περιλαμβάνεται στον κατάλογο των θεμάτων που αναφέρθηκαν προηγουμένω. Νομίζω ότι είναι η πιο σημαντική μα δράση, διότι είναι αυτή η οποία θα έχει άμεσε συνέπειε στη νέα νομοθεσία. Ευχαριστούμε για την έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, διότι μας δίνει αποδείξεις. Ε, εννοώ ότι αυτή είναι μια έκθεση που είναι αποτέλεσμα των δημοσίων ε, λειτουργών που εκφράζουν την άποψή τους και λένε ότι δεν γνωρίζουν ίσως πάρα πολλά πράγματα για το θέμα και οποιαδήποτε δράση είναι θετική. Επιβεβαιώνει λοιπόν την ανάγκη να υπάρξει ε, μία σειρά δράσεων που είναι αυτό το οποίο ε, κάναμε το Δεκέμβριο. Για μας αυτό που είναι επίσης σημαντικό είναι να υπάρχει και μία σαφής εικόνα ε, για το ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις και ποια θέματα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όταν υποστηρίζουμε τα κράτη-μέλη για θέματα παιδείας, υγείας, έλλειψης διακρίσεων, κλιμάτων μίσος και ρητορίες μίσων που είναι, μίσους που είναι όλα τμήμα των δράσεών μας γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ε, ποιε είναι οι βασικέ αρμοδιότητε των κρατών μελών σε όλου αυτού του τομεί και επομένω αυτό που κάνουμε εμεί από πλευρά μα είναι να παρέχουμε υποστήριξη σε εκείνου που θέλουν να γνωρίζουν περισσότερο επί του θέματο. Και φυσικά αυτό θα γίνει και ε, με την ε, καλύτερη κατανόηση των τομέων στου οποίου πρέπει να επικεντρωθούμε χάρη στην έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι αυτή η μάχη για να υπάρχει τελικά μια οδηγία για ε, την ίση θα προχωρήσει. Να πω ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση σαφώς και υπάρχει πολιτική, ανθρώπινη και ηθική υποχρέωση να διασφαλίσουμε την παροχή ίσων δικαιωμάτων σε όλους μας τους πολίτες. Ελπίζουμε λοιπόν κάποια στιγμή να μπορέσουμε να έχουμε ε, ένα θετικό βήμα ε, στον τομέα αυτό. Okay. As Όπως σας είπα και στην αρχή αυτής της συνεδρίασης, το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης ε, αναβάλλεται. Άρα θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και θα ξεκινήσουμε με το επόμενο σημείο σε 10 λεπτά. Στις 4 η ώρα λοιπόν φροντίστε να είστε πίσω και τώρα έχετε και λίγο χρόνο στη διάθεσή σας για ένα καφέ. So, uh, Συνάδελφοι, να ξαναξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Το επόμενο σημείο, το 7, η διάταξη, αφορά την κατάσταση στον χώρο του Σέγγεν. Νομίζω ότι όλους μας ανησυχεί η κατάσταση του χώρου Σέγγεν και τα πολυάριθμα κρατημέλη τα οποία πρόσφατα επανησύχαγαν ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα του χώρου Σέγγεν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προετοιμάσει μια ανακοίνωση με τον τίτλο «Επιστροφή στο Σέγγεν και σχετικός οδικός χάρτης» και θα πρέπει όντω να επιστρέψουμε στο Σέγγεν το οποίο γνωρίζαμε γιατί το κόστο ε, τη κατάργηση του Σέγγεν θα ήταν υπερβολικά υψηλό οικονομικό από οικονομική άποψη, αλλά κυρίω και από πολιτική άποψη. Να δώσω το λόγο λοιπόν τώρα στον κύριο Μουσέλ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας παρουσιάσει αυτή την ανακοίνωση η σύσταση της 24ης Φεβρουαρίου 2016 για τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα πρέπει να λάβει η Ελλάδα και το follow-up που έχουν λάβει τα μέτρα αυτά έως τώρα. Οι πληροφορίες που λάβαμε έως τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν για διανεμηθεί προς τα μέλη της Επιτροπής. Και μετά από την Επιτροπή θα δώσω το λόγο στην Ιλλανδική Προεδρία και τώρα ας πάρει το λόγο ο κύριος Μουσέλ. Thank you, Madam Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα αναφερθώ και στα δύο θέματα. Και την ανακοίνωση και το θέμα της Ελλάδας πολύ σωστά είπατε ότι πρέπει να επανέλθουμε στο Σέγγεν όπως το ξέραμε. Ίσως να είναι παραπλανητικός ο τίτλος. Όχι ότι δεν είμαστε πλέον στο Σέγγεν, απλά δεν λειτουργεί κανονικά το Σέγγεν αυτή την εποχή και πρέπει να επανέλθουμε στην ομαλή λειτουργία και στους, στους γνωστούς κανόνες ε, του Σέγγεν. Το Νοέμβριο του 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μια ομάδα εμπειρογνωμόνων έκανε μια επίσκεψη αξιολόγηση του Σέγγεν στην Ελλάδα που έδειξε ανεπάρκειες. Ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια ευπροηγουμενου εισρωή μεταναστών, μια γνωστό της πάση, και ο συνδυασμός αυτών οδήγησε σε πολλές δευτερογενείς μετακινήσεις που είχαν ως αποτέλεσμα την ε, θέσπιση ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα από κάποιες χώρες όπως Βέλγιο, ε, Δανία, Γερμανία, Αυστρία, Κροατία, Ελβετία, με συγγνώμη Σουηδία και Νορβηγία. Η Νορβηγία που δεν είναι βέβαια μέλος Ένωσης. Έξι από τα κράτη-μέλη εξακολουθούν τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα. Η έλλειψη στα εσωτερικά σύνορα δεν σημαίνει όμως το τέλος του Σέγγεν, αλλά ότι σε κάποια σύνορα υπάρχουν έλεγχοι σε κάποια κομμάτια των σύνορων. Και ίσως αυτό είναι το 15% των εσωτερικών σύνορων, ίσως και λιγότερο. Και δεν καλύπτουν παρά μόνο τα χερσαία σύνορα, ούτε θαλάσσια σύνορα, ούτε αέρια. Άρα για τους περισσότερους πολίτες το Σέγγεν λειτουργεί όπως πριν. Το βασικό όμως θέμα είναι ότι δεν υπήρξε συντονισμός. Εγκρίναμε λοιπόν την ανακαίνωση που λέει Back to Schengen και θέλουμε να εξασφαλίσουμε την προστασία των εξωτερικών συνόρων. Και ξέρετε ότι γι' αυτό έχουμε καταθέσει ε, μία πρόταση για την ακτοφυλακή, την αρχή για τα την ακτοφυλακή. Θέλουμε να εγκριθεί το στόμα δυνατό και από το Κοινοβούλιο για να εγκριθεί πριν το τέλος της Ολλανδικής Προεδρίας. Αυτό το πρώτο στρώμα. Το δεύτερο, να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ελλάδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι η Ελλάδα μετοπίζει μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση, όπως ξέρετε, λόγω της γεωγραφικής της θέσης. Τρίτον, Ξέρουμε ότι κάποια κράτη-μέλη διευκόλυναν τη διαμετακόμιση, τη διέλευση μεταναστών από το ένα σύνορο στο άλλο και θα πρέπει αυτή η πολιτική διέλευση, τη διαμετακόμιση να σταματήσει και σε μεγάλο βαθμό ανεκόπη με την έγκριση αυτής της ανακοίνωσης. Τέλος, η έλεγχη στα σύνορα, αν χρειαστεί να πανθυσπιστούν, θα πρέπει αυτό να γίνει με συντονισμένο τρόπο και όχι με εμβαλωματικές αποφάσεις που είχαν αυτό το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που είδαμε κατά το παρελθόν. Αυτή είναι η τέταρτη βασική άξονες της ανακοίνωσης. Αν μου επιτρέπετε τώρα θα ήθελα να τονίσω ορισμένα στοιχεία Όπως είπα, ε, κάποιες χώρες ε, διευκολύνουν τη μετακόμιση, τη διέλευση μεταναστών από το ένα σύνολο στο άλλο. Δεν είναι όμως αυτή η σωστή προσέγγιση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 18 και 19 Φεβρουαρίου ανέφερε ξεκάθαρα ότι αυτή δεν είναι από νομικής πλευράς η ορθή προσέγγιση. Το Δουβλίνο επίση πρέπει να εφαρμοστεί. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος ετηθεί άσυλο και ήταν σε ένα κράτος μέλος πριν, θα πρέπει να σταλεί στο πρώτο. Μπορεί να μην σας αρέσει το Δουβλίνο σε όλους και επεξεργαζόμαστε μια μεταρρύθμιση αυτής της συνθήκης και θα την έχετε ε, τη σχετική πρόταση, αλλά προτού έχουμε ένα καλύτερο σύστημα πρέπει να εφαρμόσουμε το ισχύον. Αυτό σημαίνει ότι και η Ελλάδα πρέπει να εφαρμόσει το σύστημα αυτό, πρέπει να εφαρμόσει το Δουβλίνο γιατί οι μετανάστες ήξεραν ότι μπορούσαν να συνεχίσουν και δεν θα στέλνονταν πίσω στην Ελλάδα. Και ήταν εκτός Δουβλίνου η Ελλάδα. Θέλουμε λοιπόν να δούμε το ενδεχόμενο να ξαναμπεί μέχρι τον Ιούνιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου, η Ελλάδα πίσω στο Δουβλίνο και εμείς θα αξιολογήσουμε το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν μέχρι τον Ιούνιο μεταφορές στην δυνάμει του Δουβλίνου. Ώστε τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τους κανόνες του Δουβλίνου. Και αυτό θα περιορίσει και αυτές τις μετακινήσεις. Τι θα πει να εξασφαλίσουμε τη συντονισμένη προσέγγιση. Ξέρετε ότι υπάρχει δυνατότητα επανεισαγωγή συνοριακών ελέγχων για δύο μήνες. Και αυτό σε περίπτωση κατεπήγοντος, όταν δηλαδή απαιτείται κατεπήγουσα δράση. Υπάρχει και μια άλλη δυνατότητα. Το άρθρο 25. Για έξι μήνες σε περίπτωση σοβαρής απειλή για τι δημόσιες πολιτικές στην εσωτερική ασφάλεια. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ιδιαίτερω ευέλικτοι. Αφήσαμε τα κράτη-μέλη να μπορούν να, να επαναθεσπίσουν για 8 μήνες του συνολικού ελέγχου. Έξι και 2. Δηλαδή συνδυάσαμε τα άρθρα 23 και 25. Όμως τώρα για τη Γερμανία λίγη η περίοδος τέλη Μαΐου, μέχρι τις 30 Μαΐου δηλαδή, μετά τις 30 Μαΐου, δεν θα υπάρχει νομικό πλαίσιο που να επιτρέψει τη Γερμανία να συνεχίσει τους έλεγχους εσωτερικά τη σύνορα και για κάποια άλλο όπως η Αυστρία θα έχουμε άλλες προθεσμίες όπως είναι 16 Μαΐου για την Αυστρία και άλλα κράτη πιο αργά. Πρέπει να βρούμε μια προσέγγιση όμως για το τι θα ισχύσει μετά τις 30 Μαΐου. Και αυτό μας απασχολεί λοιπόν στην ανακοίνωσή μας. Και τώρα έρχομαι στο δεύτερο θέμα που είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Όπως γνωρίζετε, Το Νοέμβριο του 2015 έγινε μια επίσκεψη στην Ελλάδα, όπου εντοπίσαμε σοβαρές ανεπάρκειες στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων από την Ελλάδα. Αυτό ως αποτέλεσμα μια εφαρμοστική απόφαση από το Συμβούλιο με συστάσεις συγκεκριμένες προς την Ελλάδα για να διορθώσει τις ανεπάρκειες. Αυτή λοιπόν η εφαρμοστική απόφαση δημοσιοποιήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου. Δύο εβδομάδες μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντενέκρινε μια εφαρμοστική απόφαση που ρύθμιζε ε, τα ειδικά μέτρα που πρέπει να λάβει η Ελλάδα υπομορφήν σύστασης για να συμμορφωθεί προς τις ε, συστάσεις του Συμβουλίου. Είναι λίγο πολύ, προκαλεί καταλαβαίνετε. Πρώτα αντέδρασε το Συμβούλιο, μετά η Κομισιόν κτλ. Μετά τι συστάσει και Συμβουλίου και Κομισιόν, η Ελλάδα κοινοποίησε ένα σχέδιο δράση, το οποίο αναφερθήκατε και εσείς, γιατί απεστάλληκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα, συγκεκριμένα στις 17 Μαρτίου, Και τώρα έχουμε ένα σχέδιο δράσης από την Ελλάδα για να διορθωθούν αυτές οι ανεπάρκειες, όπως είπα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή, την ώρα που μιλάμε, αξιολογεί αυτό το σχέδιο δράσης. Έχουμε ένα μήνα στη διάθεσή μας. Μέχρι τις 12 Απριλίου πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει την αξιολόγηση και το αργότερο τότε θα διαβιβάσουμε στο Συμβούλιο την αξιολόγησή μας. Ερχόμαστε σε επαφή και με τους εμπειρογνώμονες, οι οποίοι κάνουν και αυτοί που έκανε την αξιολόγηση ε, τον Νοέμβριο του 2015, την αξιολόγηση για το Σέγγεν. Και όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, και πριν ολοκληρωθεί βέβαια δεν μπορώ να σας πω τίποτε πιο αναλυτικό για αυτή την αξιολόγηση, αφού μόλις λάβαμε το έγγραφο. Όταν όμως περάσουν τρεις μήνες από την αξιολόγηση, δηλαδή μέχρι τις 12 Μαΐου του 2016, η Ελλάδα θα αναφέρει σε ό,τι αφορά την εφαρμογή αυτών των συστάσεων. Και τότε θα μπορούμε, δηλαδή μέχρι τις 12 Μαΐου επαναλαμβάνω, να αποφασίσουμε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Και μια από τις επιλογές είναι η έγκριση μιας πρότασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρόταση σύστασης, δυνάμει το άρθρο 26 παράγραφος 2 του κώδικα για τα σύνορα του Σέγγεν, είναι όμως η έσχατη λύση. Και με ένα τέτοιο μέτρο από κοινού και με συντονισμένο τρόπο θα μπορούμε να διατηρήσουμε κάποιου έλεγχου αστερικά σύνορα ήδη εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για να διορθωθεί η κατάσταση. 26 παράγραφος 2, 26 άρθρο παράγραφος 2 λοιπόν. Αλλά μόνο για δύο χρόνια ε, μπορεί να ισχύει η επανεισαγωγή των ελέγχων. Δεν λέω ότι θα γίνει, λέω ότι αξιολογούμε την κατάσταση και θα δούμε αν χρειαστεί να γίνει όχι. Και σε κάθε περίπτωση τονίζω ότι αν γίνει θα είναι για να διορθωθεί η κατάσταση. Και μιλάμε για συγκεκριμένους ε, συνορικούς σταθμούς. Δεν σημαίνει ότι θα έχουμε συνορικούς ελέγχους για όλες τις μεταφορές χερσαίες, εναέριες θαλάσσιες. Μπορεί να είναι περιορισμένο για κάποιες χερσαίες για κάποια χερσαία σύνορα, συγκεκριμένε περιοχέ. Άρα να γίνει κατανοητό παρακαλώ ότι στόχο μα είναι να δοθεί μια συντονισμένη ανταπόκριση σε περίπτωση που εξακολουθεί να είναι αναγκαία η εφαρμογή συνοριακών ελέγχων στα αστερικά σύνορα. Ο στόχο μα όμω είναι, όπω είπα, η ομαλοποίηση, να επανέλθουμε στην ομαλή λειτουργία του Σέγγεν και τα κράτη-μέλη όλα μαζί ομοιόμορφα και συλλογικά κινούνται. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την έκθεση αυτή, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χαίρομαι που έχουμε πλέον και γραπτές πληροφορίες για την αξιολόγηση του χώρου Σέγγεν και φυσικά τις συστάσεις ε, που προκύπτουν από τις ε, γραπτές αυτές παρατηρήσεις. Ε, πριν δώσω το λόγο στο Συμβούλιο για να μας μιλήσει για τις στάσεις ε, της 12 Φεβρουαρίου του 2016 προς την Ελλάδα για να μειώσει τις ανεπάρκειες, να σας πω επίσης ότι σήμερα υπάρχει εκπρόσωπος της μόνιμης αντιπροσωπείας της Ελλάδος εδώ και επομένως ε, θα ήταν χρήσιμο να έχουμε και κάποιες απόψεις εκ των έσω, απευθείας από την Ελλάδα. Πρώτα όμως να δώσω το λόγο στο Συμβούλιο στον κύριο Λούστεμπορκ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο για να σας μιλήσω για τη σύσταση του Συμβουλίου της 12 η Φεβρουαρίου. Πρόκειται λοιπόν για εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου που ε, κάνει συστάσεις προς την Ελλάδα. Πρόκειται για μια σύσταση η οποία εγκρίθηκε βάσει της νέας αξιολόγησης Σέγγεν του κανονισμού του 2013 και βάσει αυτού του κανονισμού το Συμβούλιο εγκρίνει κατόπιν πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συστάσεις προς τα κράτη-μέλη προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ανεπάρκειες που εντοπίστηκαν κατά την αξιολόγηση Σέγγεν. Στη σύσταση αυτή προς την Ελλάδα λοιπόν δεν έχουμε την πρώτη ε, σύσταση, έχουμε αρκετές συστάσεις από τότε που ξεκίνησε ο πρώτος μηχανισμός εξολόγησης στη λειτουργία του. Οι συστάσεις αυτές βασίζονται λοιπόν στις τελικές εκθέσεις οι οποίες ε, συζητούνται και αποφασίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βασίζονται στις επιτόπιες ε, επισκέπτες που γίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Το Νοέμβριο έγινε και σχετική επίσκεψη στην Ελλάδα. Ε, οι συγκεκριμένε συστάσεις λοιπόν για την Ελλάδα αποτελούν συνέχεια της ευνηδιαστικής επίσκεψης που έγινε το Νοέμβριο και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βασίστηκε σε αυτή την τελική έκθεση που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 2 Φεβρουαρίου. Επειδή είναι κατεπήγον ο χαρακτήρας της ε, στην Ελλάδα και ε, επειδή η φύση των ε, ανεπαρκειών είναι συγκεκριμένη, το Συμβούλιο συνεργάστηκε πολύ στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ελλάδα προκειμένου να εγκρίνει αυτές τις στάσεις το συντομότερο δυνατόν και το Συμβούλιο τις ενέκρινε στις 12 Φεβρουαρίου. Οι συστάσεις αυτές επικεντρώνονται στα στοιχεία τα οποία προέκυψαν από τις ε, επισκέψεις, παραδείγματο χάρη τη διαδικασία καταγραφής, αναγνώρισης ταυτότητας και παρακολούθησης. Η Ελλάδα τώρα εργάζεται πολύ σκληρά για την εφαρμογή των συστάσεων και όπως είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Ελλάδα ε, ε, έχει πλέον ένα σχέδιο δράσης το οποίο ε, ανακοίνωσε και στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το επόμενο βήμα αυτής της διαδικασίας όπως εξήγησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι κάτι το οποίο αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σαφέστατα και ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα αξιολογεί το ελληνικό σχέδιο δράσης, το Συμβούλιο πρέπει να περιμένει την αξιολόγηση και από εκεί και πέρα η Ελλάδα θα πρέπει ε, να φροντίσει να εφαρμόσει το σχέδιο δράσης μπορεί να επανέλθει το θέμα στο Συμβούλιο, αλλά προς το παρόν το Συμβούλιο περιμένει την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα αποτελέσματα της ε, ελληνικής εφαρμογής του σχεδίου δράση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τις απόψεις σας και τις ε, συστάσεις του Συμβουλίου. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Βούλγαρη από την ε, μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδος, έχετε κατά νου ότι οτιδήποτε αποφασίζεται στον χώρο Σέγγεν δεδομένου ότι έγινε και μόλις ε, πρόσφατα μια ψηφοφορία στην Επιτροπή μας ε, για την ολιστική προσέγγιση για τη μετανάστευση. Πρέπει λοιπόν να έχουμε κατά νου ότι για να υπάρξουν αποτελέσματα σε ένα τομέα πρέπει να ε, υπάρξουν αποτελέσματα και στους άλλους τομείς της μετανάστευσης. Αυτό είναι σημαντικό να το ξέρουμε γιατί δεν υπάρχει μία απάντηση για τη μετανάστευση. Να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Βούλγαρη πριν δώσω το λόγο στους συναδέλφους και σας παρακαλώ όσοι θέλετε να σχολιάσετε να μου το πείτε. Κύριε Βούλγαρη, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Όπως ευκρίνησε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μία ε, ε, ευνηδιαστική ε, επίσκεψη έλαβε χώρα στην Ελλάδα, στα σύνορα με την Τουρκία, τον Νοέμβριο του περσινού έτους. Και η επίσκεψη αυτή κάλυψε τη Σάμο, και τα σημεία στις ε, Καστανιές, ε, ε, Οριστιάδα και Φυλάκιο Ήταν τεράστιες οι δυσκολίες λοιπόν σε ό,τι αφορά την άνευ προηγουμένου κρίση προσφύγων. Είναι α, χωρίς προηγούμενο αυτές οι καταστάσεις. Υπάρχει ένα πρόβλημα με το μικρόφωνο του ομιλητή. Αν θα μπορούσατε να αλλάξετε μικρόφωνο γιατί δεν ακούν καλά οι διερμηνείς. Ένα πρόβλημα με το μικρόφωνο σας παρακαλώ αλλάξτε θέση, αλλάξτε μικρόφωνο γιατί δημιουργείται πρόβλημα. Σας ζητώ συγγνώμη. Ελπίζω να δουλέψει καλύτερα βεβαίως. Ναι. Το μικρόφωνο του μιλητή λειτουργεί εξαιρετικά. Μάλιστα. Σας μιλούσα λοιπόν για την επίσκεψη που έλαβε χώρα στα διάφορα νησιά, στα νησί της Σάμου, της Χίου και στο σημείο ε, Νεοφυλάκιο Καστανιάς Ορτιάμπα και Νέα Βίζα. Όλοι αναγνωρίζουν τις ιδιαίτερες δυσκολίες που ε, συνεπάγεται η αντιμετώπιση αυτής της κρίσης ε, μεταναστών άνευ προηγουμένου οι εκτάσεις της και ιδιαίτερα οφείλεται αυτό στην Ελλάδα λόγω της, στη γεωγραφική της θέση και έτσι αυτής η ένταση, αυτής η διάστασης ε, κρίση θα σήμαινε πίεση για όλα τα κράτη-μέλη Όλοι ξέρουμε ότι βασικός μας στόχο είναι να σεβαστούμε το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο και να σώσουμε ανθρώπινε ζωέ και να εφαρμόσουμε στην πράξη τις ευρωπαϊκές ανθρωπιστικές μα αξίε. Είναι μεγάλη πρόκληση και δύσκολη δουλειά. Οι, ευρωπαϊ... οι αρχές κατέφεραν να σώσουν πάνω από 100.000 πρόσφυγες και μετανάστες άτομα σε κατάσταση έκτακτη ανάγκη από πέρσι σε πολλά τέτοια περιστατικά. Η Ελλάδα θεωρεί κάθε σεβασμό ότι τα ευρήματα της αξιολόγησης δεν λαμβάνει υπόψη τα σοβαρά προβλήματα και δεν δείχνουν, ε, δεν αποδεικνύουν ότι η, η Ελλάδα η Ελλάδα αμέλησε τις υποχρεώσεις της και δεν ε, καταλαβαίνουν το τι σημαίνει αυτό για άλλα τα κρατη Έχουν σημειωθεί πολλοί πρόοδοι για να, για να καλυφθούν τα κενά που έχουν εντοπίσει αξιογοι ελογήσεις ακόμα και πριν τις την 25η Φεβρουαρίου με τις συστάσεις του Συμβουλίου και της ε, Επιτροπής 24 Φεβρουαρίου η, Ευρω... η Ελλάδα συνεργάζεται στενά με όλες τις υπηρεσίες και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με άλλα κράτη-μέλη για να ανταποκριθεί σε αυτές τις μεγάλες και δυσανάλογες μεταναστευτικές πιέσεις και έχουν κινητοποιηθεί όλοι οι πόροι που έχουμε στη διάθεσή μας. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, ακόμα και πριν την συστάσεις, οι ελληνικές αρχές προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν τα κενά που υπάρχουν. Μετά την έκδοση των συστάσεων, όπως είπε η Προεδρία, κάναμε τα απαραίτητα βήματα και καταρτήσαμε ένα σχετικό σχέδιο δράση στις 12 Μαρτίου σε στενή συνεργασία με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου δράση αυτού. Πολλές ενέργειες έχουν ήδη ολοκληρωθεί, για παράδειγμα στο θέμα της καταχώρησης και σε ό,τι αφορά την διεξαγωγή των ε, συνοριακών ε, ε, διαδικασιών. Αυτό προαπαιτεί προσπάθειες από όλους και όχι μόνο από την Ελλάδα. Συλλογικά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις σε ένα πνεύμα κοινή ευθύνη και αλληλεγγύης. Δεν είναι η κρίση της Ελλάδας, δεν είναι η κρίση της Ευρώπης αυτής. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ακούσαμε λοιπόν τρεις διαφορετικές απόψεις. Ίσως να υπάρχουν κάποιες συγκλήσεις απόψεων φυσικά για τα θέματα αυτά, αλλά ευχαρίστω να δώσω το λόγο και σε όλους τους συναδέλφους που τον έχουν ζητήσει. Η κυρία Έρνης ήταν η πρώτη που ζήτησε το λόγο. Ναι, ήθελα να έχω λίγο χρόνο να ηρεμήσω, αλλά να πάρω το λόγο πρώτη. Σε ό,τι αφορά την παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να σας πω ότι θα πρέπει να σταματήσει η πολιτική που ασκείται σε ό,τι αφορά αυτή την πολιτική που τι σημαίνει ότι οι άνθρωποι που θέλουν άσυλο δεν τους δίνεται η ευκαιρία να κάνουν ε, το αίτημα αυτό και όλη η Επιτροπή ουσιαστικά προσφύγων στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε Σε ό,τι αφορά την Τουρκία τώρα, Ό,τι συμβαίνει ουσιαστικά παραβιάζεται η συνθήκη της Γενέβης. Πώς το συνδυάζεται λοιπόν αυτό σε αυτή την πολιτική του πασαρίσματος, της προώθησης των ετούντων ασύλο. Πώς συνδυάζεται αυτό με την συνθήκη της Γενέβης και ότι έχει απομείνει από αυτήν. Είπατε ότι θα πρέπει να τηρήσουμε το Δουβλίνο. Και θα πρέπει να κοιτάξει η Ελλάδα μέχρι τον Ιούνιο πώς μπορεί να εφαρμόσει καλύτερα το, τη συνθήκη του Δουβλίνου. Να σας πω ειλικρινά, στο Φεβρουάριο, μέσα το Φεβρουάριο, στην Ελλάδα ήταν 868.000 τα άτομα που καταφτάσαν στην Ελλάδα για να περάσουν στην Ευρώπη. Σήμερα το πρωί λοιπόν τα στοιχεία ήταν 50.411 άτομα τα οποία έχουν προσταθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Μιλάμε σχετικά, σχετικά για ένα εκατομμύριο δηλαδή άτομα τα οποία καταφθάνουν στην Ελλάδα για να προωθηθούν στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν πρόκειται να σταματήσουν οι ροές αυτές. Μα πώς δηλαδή φαντάζεστε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να τηρήσει το Δουβλίνο. Είναι πραγματικά ένιγμα αυτό για μένα. Πώς το εννοείτε. Θεωρώ ότι είναι τελείως αντιπαραγωγικό αυτό. Και όλοι σας το ξέρετε, το ξέρετε και το ξέρετε 100% ότι έχει αποτύχει το Δουβλίνο και δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Σε όλα αυτά που λέτε για τα εσωτερικά σύνορα, για τα εξωτερικά σύνορα, για το Σέγγεν, λείπει, λείπει το στοιχείο της κριτικής προς τα κράτη-μέλη, τα οποία με την πολιτική τους οδηγούν να κάθονται και να περιμένουν χιλιάδες άτομα στα εσωτερικά σύνορα, της Ευρώπης και ότι εισαγάγονται συνοριακοί έλεγχοι, δηλαδή για οκτώ μήνες οι οποίοι έχουν περάσει για τη Γερμανία θα πρέπει να βρούμε κάτι άλλο τώρα και το Σέγγεν κλειδονίζεται στο μεταξύ. Ε, κάντε κριτική στην Ελλάδα, μα θέλετε, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά δεν γίνεται. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω και την ε, άποψή σας για την ιστορία αυτή για τα ιστορικά σύνορο. και για τα εξωτερικά σύνορα και την προστασία τους από τους ε, πρόσφυγες. Μπορούμε να φροντίσουμε ότι θα υπάρχει καλύτερη καταχώρηση των προσφύγων στα σύνορα. Ακούσαμε τέτοια και την προηγούμενη εβδομάδα. Το καταλαβαίνω αυτό. Είναι σωστό. Αλλά τι να κάνουμε δηλαδή. Pushback. Ξέρουμε ότι απαγορεύεται Είμαι κοινική Ελλάδα, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Η Ελλάδα σύστασε 34 κέντρα υποδοχής, τα οποία είναι πραγματικά ε, τελείως γεμάτα πλέον. Και ουσιαστικά τίποτα δεν έχει περάσει στην κεντρική Ευρώπη. Και ουσιαστικά μία ρύθμιση που πετύχαμε για την Τουρκία, η οποία και αυτή για γέλια είναι, αν είμαστε κοινικοί. Είναι πραγματικά γελία η κατάσταση και αυτά που μας ε, σερβίρεται σήμερα. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να γελάσω κοινικά και το θεωρώ επονίδιστο. Έχετε πάει ποτέ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Συμβούλιο εκεί να δείτε τι γίνεται στα σύνορα. Να δείτε τι διαμείβεται. Αν θέλετε να πάω εγώ μαζί σας. Να έρθω εγώ μαζί σας, γιατί θα το κάνουμε και από πλευρά της ομάδας μου σύντομα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και η Πρόεδρος. Μια και δεν είναι όλα τα μέλη εδώ, δεν ήθελα να περιορίσω τον χρόνο ομίλιας των συναδέλφων. Άλλοι τέσσερις συνάδελφοι προς το παρόν είναι στον κατάλογο. Πέντε, πέντε συνάδελφοι είναι στον κατάλογο των ομιλητών. Να ολοκληρώσουμε μέχρι τις 5.30. Έχουμε χρόνο, αλλά σας παρακαλώ μην μακρηγορείτε ιδιαίτερα. Ο κύριος Ντεπρέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να ζητήσω συγγνώμη που έφτασα λίγο αργά, άρα κάποια από τα ερωτήματά μου ενδεχομένως να έχουν ήδη απαντηθεί. Καταρχάς θέλω να πω ότι είμαι υπέρμαχος του Σέγγεν ανεφόρων, θεωρώ ότι είναι ένα από τα δομικά και εκτιμένα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και δεν ήταν καταστροφικό να πάψει να ισχύει. Χαίρομαι λοιπόν που είχαμε αυτή την ανακοίνωση με την οποία ορίζονται τα στάδια για την επανοικοδόμηση του χώρου Σέγγεν. Τούτου λεχθέντος όμως. Έχω κάποιες ερωτήσεις σε ό,τι αφορά την Ελλάδα. Βλέπω εδώ το χρονοδιάγραμμα. Σε ένα σημείωμα για αυτό το back του Schengen. Για τις 16 Μαρτίου βλέπω εδώ ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τροποποίηση του κανονισμού του Δουβλίνου βάσει της αρχής της αλληλεγγύης και της ισομέρους κατανομής των βαρών μεταξύ των κρατών μελών. Μπορεί να μην πρόσεχα και πολύ, αλλά μου ξέφυγε, δεν ξέρω, δεν το έχω πάντως ε, προσέξει να είναι μέσα στην ανακοίνωση Κομισιόν αυτό. Υπάρχει, θα μας ανακοινωθεί. Αλλά δεν είναι αυτή η ουσία της παρέμβασής μου. Το λοιπόν, 16 Μαρτίου θα έχουμε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής για την αναθεώρηση. Μεταρρύθμιση. Τον Ιούνιο όμως θα παρουσιάσει την αξιολόγησή της για ενδεχόμενη επανάληψη των ε, κινήσεων των μεταφορών στην Ελλάδα με δυνάμει του κανονισμού του Δουβλίνου, του προηγούμενου κανονισμού υποθέτω, έτσι. Τι είναι αυτό το χρονοδιάγραμμα. Προτείνουμε πρώτα μεταρρύθμιση ή τροποποίηση και μετά λέμε επανέρχεται ο κανονισμός ο ίδιος που θέλουμε να τροποποιήσουμε. Ή το πάντων δεν κατάλαβα τίποτα. Και όπως και αν έχει με εκπλήσει το αδιέξοδο που αυτή τη στιγμή ε, υπάρχει στην Ελλάδα. Δηλαδή φτάνουν ε, οι μετανάστες, δεν υπάρχει δυνατότητα να φύγουν. Η Βουλγαρία κλείσε, η Μακεδονία κλείσε, η Αλβανία μάλλον θα τα κλείσει αν δεν τα έχει δικλείσει. Άρα έχουμε ήδη δεκάδες χιλιάδες άτομα ε, στην Ελλάδα που είναι αποκλεισμένα εκεί πολύ αισιόδοξα τα βλέπει η Κομισιόν που λέει ότι με τα μέτρα που θα ληφθούν με την Τουρκία θα μειωθεί γρήγορα ο αριθμός των αφήξεων στην Ελλάδα. Και για να αντισταθμιστεί μάλλον αυτός ο αριθμός θα παναπατριστούν αυτοί οι οποίοι είχαν περάσει από την Ελλάδα και πήγαν κάπου αλλού, μα με βάση ποια κριτήρια. Ένα εκατομμύριο είναι στη Γερμανία. Τέλο πάντων, τα λέω γιατί προσπαθώ να καταλάβω, κύριοι. μην περνάτε από την Ελλάδα, ε, γυρίστε πίσω, γιατί πάλι θα σε... Δεν καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω τη λογική. Ούτε αυτό το μηχανισμό τον καταλαβαίνω. Είναι ψευής πόθη. Αφήστε που θα δημιουργήσει μια κατάσταση που θα μπορούμε να τη διαχειριστούμε. Έχετε δει ε, στα σύνορα με τη Μακεδονία αυτές τις επονίδιστες εικόνες από τους καταβλισμούς. Πώς μπορούμε πολιτισμένοι άνθρωποι όπως εμείς να αφήνουμε σε απόγνωση αυτούς τους ανθρώπους σε αυτή την κατάσταση. Ανθρώπους που είναι ήδη απελπισμένοι. και θα δώσουμε κάποια εκατομμύρια στην Ελλάδα για να τους υποδεχθεί. Ωραία, θα γυρίσουν πίσω ένα εκατομμύριο, όχι. Πώς θα γυρίσουν πίσω με αυτόν τον κανονισμό. Και ποιος θα επιλεγεί, πότε, από ποια χώρα. Συγγνώμη, αλλά ειλικρινά τα διαβάζω και δεν τα πιστεύω αυτά που βλέπω μπροστά μου. Στο πολύ κύριε Βουλευτή, επόμενος, επόμενη κυρία Στίβενς και μετά κύριος Κοέλιο. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε και συνάδελφοι. Χαίρομαι που λάβαμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ε, επιστροφή στην κανονική λειτουργία του ΣΕΝΙΑ. Θα πρέπει φυσικά να λάβουμε υπόψη και την κατάσταση στα κράτη-μέλη. Κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν μαζική εισρωή προσφύγων. Αλλά πιστεύω ότι η Ευρώπη θέλει να επιτύξει αλληλεγγύη. Αλλά όπως δικαίως επεσήμωνε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ασφάλεια και η προστασία των εξωτερικών σύνορων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα πρέπει δικαίως να αποτελεί κοινή ευθύνη και όλοι θα πρέπει να λάβουν τις ευθύνες τους σε πρώτη φάση σε επίπεδο κρατών μελών. Φυσικά όμως θα πρέπει τα κράτη-μέλη να τα βοηθήσει σε περίπτωση που χρειάζεται και η Frontex και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να ζητούν και αυτά Άρα Η εθνική υπερηφάνεια δεν θα πρέπει να εμποδίζει και το αίτημα για βοήθεια, γιατί αυτό συνέβη τους τελευταίους μήνες και είναι πραγματικά κρίμα. Η συμφωνία με την Τουρκία αναφέρθηκε ήδη πολλάκις στη συζήτηση. Η συμφωνία προέκυψε γιατί τα κράτη-μέλη δεν έκαναν ό,τι έπρεπε να έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια και ως εκ τούτου βρισκόμαστε σήμερα σε μια δύσκολη κατάσταση και φυσικά η Τουρκία θα αποφεληθεί, θα προσπαθήσει να αποφεληθεί από την κατάσταση αυτή. Εμείς θα πρέπει να φροντίσουμε να τηρήσει το δικό της σκέλος της συμφωνίας η Τουρκία και θέλω να τονίσω ιδιαίτερος ότι θα πρέπει σε ό,τι αφορά το, τους πρόσφυγες και τους μετανάστες θα πρέπει να μπορούν να περάσουν στη χώρα στην οποία επιθυμούν να βρίσκονται. Θα πρέπει όμως να τονίσουμε ότι θα πρέπει να ελέγχονται όλοι οι μετανάστες, οι πρόσφυγες στα εξωτερικά σύνορα. Και θα πρέπει να εφαρμοστούν πλήρως ε, τα όσα προβλέπει το Δουβλίνο. Ο συναδέλφος Ντεπρέ αναρωτιέται τι συμβαίνει με τους ε, πρόσφυγες που ήδη έχουν μπει στην Ένωση, αλλά νομίζω ότι η συμφωνία με την Τουρκία ισχύει μόνο για τους πρόσφυγες που θα έλθουν ε, και θα καταφτάσουν από εδώ και πέρα, από σήμερα και πέρα. Όχι για όσους ήδη έχουν καταφτάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τι γίνεται με τους πρόσφυγες που βρίσκονται στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στο Βέλγιο θα πρέπει να ξαναεπιστραφούν στην Ελλάδα. Θα πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό προσεκτικά, γιατί η Ελλάδα αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα με του ανθρώπου που έχει εκεί. Αυτό εξαρτάται ασφαλώ και από την κατάσταση στην Ελλάδα την ίδια. Και με χαρά άκουσα το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τα άτομα τα οποία έρχονται από τρίτες χώρες δεν μπορούν να έχουν πλέον πρόσβαση στην Ευρώπη αν δεν έχουν καταθέσει έτοιμα για θεώρηση για να έχουν ζητήσει άσυλο στα εξωτερικά σύνορα. Αυτό μου φαίνεται πραγματικά προφανές. Αυτό σημαίνει ότι επιτέλους ε, χρησιμοποιούμε και λίγο την κοινή μας λογική. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Ο συνοριακός ε, κώδικας του Σέγγεν δεν είναι μόνο έτσι ένα απλό έγγραφο και το έλεγα πάντα ότι όσο ισχύουν οι κανόνες του Δουβλίνου θα πρέπει να ισχύουν. Γιατί οι κανόνες είναι κανόνες. Μας αρέσουν, δεν μας αρέσουν, θα πρέπει να ισχύουν. Και αν υπάρχει επιβαλλική επιβάρυνση σε χώρες θα πρέπει να ζητούν βοήθεια. Όχι απλά να προωθούν τον κόσμο και να προωθούν και τα προβλήματα μαζί με τον κόσμο αυτό. Γιατί αυτή η αντιμετώπιση είναι που μας έχει προκαλέσει τα σημερινά προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κοέλιο και μετά η κυρία Βεριζιά. Κύριε Κοέλιο, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω δύο λόγια αντίστοιχα με αυτά του κυρίου Ντεπρέ. Και εγώ είμαι υπέρμαχος ε, της Σέγγεν και πιστεύω ότι η προτεραιότητά μας αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι η προστασία της Σέγγεν. Όπερ και πρέπει ο όρος αλληλεγγύη να γίνει πράξη. Να υπάρξει μεγαλύτερο συντονισμός, ε, μικρότερες καταχρήσεις των εθνικών καταστάσεων, μια συνολικότερη προσέγγιση και να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε μέτρα ε, τα οποία ε, είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση αυτή του οδικού της χάρτη η οποία ε, παρεπιπτόντως ε, μας λέει ότι ε, θέλει να αξιολογήσει πλήρως το μηχανισμό Σέγγεν. Ο μηχανισμός της Σέγγεν δεν είναι μόνο η προστασία των συνόρων, αλλά μια σειρά από μέτρα που εγγυώνται την καλή λειτουργία Σέγγεν. Παραδείγματος χάρη ο μηχανισμός αξιολόγησης της Σέγγεν και στον οποίο επιμένετε στον οδικό σας χάρτη. Δεν θα αναφερθώ στην Τουρκία, δεν είναι ακόμα η στιγμή να εκφράσουμε τις επιφυλάξεις μας επί του θέματος, αλλά όσον αφορά αφορά την Ελλάδα, ε, συμφωνώ απολύτως με την ιδέα ότι τα διαρθρωτικά προβλήματα της Ελλάδος χρήζουν λύσεις μεν, αλλά υπάρχουν και κάποια συγκυριακά προβλήματα τα οποία απορρέουν από αυτή την μαζική αύξηση, ε, άφηξη ανθρώπων. Οι ευνηδιαστικές επισκέψεις στην Ελλάδα αποδεικνύουν πραγματικά ότι η Σέγγεν διαθέτει τα εφόδια για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα, αλλά ε, σας ευχηστώ την προσοχή, αυτό δεν αρκεί για να επιληθούν τα προβλήματα της Ελλάδος. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ροή ανθρώπων και υπάρχουν και διαρθρωτικά προβλήματα. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ολοκληρώσω με αυτό το οποίο με ανησυχεί περισσότερο στον οδικό χάρτη. Το άρθρο 26 και η δυνατότητα παράτασης κατά δύο χρόνια των εσωτερικών ελέγχων στα σύνορα. Δεν θα ήθελα τώρα να ε, σας αναπτύξω εδώ όλα τα ερωτηματικά που μου τίθενται όσον αφορά την νομιμότητα αυτής της ε, πρότασης. Τα όσα προβλέπονται στη Σέγγεν δεν είναι λευκή επιταγή προς τα κράτη-μέλη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε καμία περίπτωση. Και επομένως θα ήθελα να πιστέψω ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ θα ελέγξουν πάρα πολύ σοβαρά το μηχανισμό πραγματικά αμφιβάλλω κατά πόσον θα μπορέσουμε ε, να αποδεχτούμε τη χρήση αυτού του μέτρου απλώς ε, λόγω των μεγάλων μεταναστευτικών πιέσεων. Σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτό το πνεύμα του άρθρου και δεν θα πρέπει ε, να το ερμηνεύσουμε έτσι επειδή δεχτήκαμε σε μια αξιολόγηση Σέγγεν ε, ότι μπορεί σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις να επανέρχονται οι έλεγχοι στα σύνορα και να μπορούν να ισχύουν και για δύο χρόνια. Ε, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι η Σέγγεν αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ευρωπαϊκού οράματος, επομένως αν θέλουμε πραγματικά ε, να το τηρήσουμε αυτό θα πρέπει η Σέγγεν να επανέλθει στην πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να επανέλθει ομαλότητα και πρέπει να προστατεύσουμε τη Σέγγεν, αλλά προφανώς ε, υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις για το πώς μπορεί να υλοποιηθεί αυτό. Η κυρία Βερζιά στη συνέχεια και μετά η κυρία Γκόμες. Νομίζω ότι έχετε δίκιο κυρία Πρόεδρε. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι ε, για να τα εφαρμόσουμε και ορισμένε φορέ αναρωτιέμαι τι ακριβώ συζητούμε εδώ. Λέμε ότι πρέπει να περιορίσουμε την μεταναστευτική κρίση. Κανένα κράτος μέλος δεν έχει ζήσει αντίστοιχε μεταναστευτικές ε, πιέσει, Είναι δυσανάλλαγη η μεταναστευτική πίεση. Να σα υπενθυμίσω τα στοιχεία. 850.000 άνθρωποι αφήχθησαν στην Ελλάδα βάσει των ε, διεθνών στοιχείων μετανάστευσης, το 80% αυτών των ανθρώπων είναι πρόσφυγες. 80-85% πρόσφυγες βάσει διεθνών οργανισμών που ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Τι κάνουμε λοιπόν. Φαίνεται ότι θέλουμε να σεβαστούμε τη διεθνή νομοθεσία και να σώσουμε ζωές. 3.770 νεκροί στη Μεσόγειο. Ανήκουστος αριθμός. Και πραγματικά τι κάνουμε εμείς για την αλληλεγγύη. Θα στείλουμε επιπλέον αστυνομία στην Ελλάδα. Ε, συγγνώμη, αλλά πραγματικά είμαι ιδιαίτερα επιφυλακτική και νομίζω ότι κάπου χρησιμοποιούμε μια ορολογία εντελώς αντιφατική. Θυμάμαι ότι μετά από αυτή την ε, περιβόητη έκτακτη σύνοδο κορυφής που ήταν έκτακτη μόνο κατόνομα τον Απρίλιο ε, στην οποία για πρώτη φορά ε, συζητήθηκε το θέμα, έγινε μετά, συγγνώμη, από την, ε, το ναυάγιο στη Λιβύη, ε, ε, μεταξύ Λιβύης και Ιταλίας και αποφάσισαν να αναθεωρήσουμε το θεματολόγιο για τη μετανάστευση. Σε αυτό το θεματολόγιο υπάρχει ένα θέμα το οποίο δεν ανάφερε ποτέ το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η νόμιμη οδοί μετανάστευσης αν δεν ανοίξουμε νόμιμες οδούς μετανάστευσης, αν δεν υπάρχουν προστατευμένοι διάβλοι για τους ε, πρόσφυγες, όχι μόνο δεν κάνουμε τίποτα, αλλά ουσιαστικά τους πρόσφυγες τους στέλνουμε σε ολοένα και πιο θανατηφόρες οδούς θα περάσουν από αλλού, θα αποφύγουν να ε, κάνουν οτιδήποτε. Ξέρουν όλοι ότι όσο περισσότερα σύνορα κλείνουμε, τόσο περισσότερους νεκρούς αφήνουμε. Διότι θα αφήσουμε στους διακινητές να ε, κάνουν φρικαλαιότητες και πραγματικά η Ελλάδα πρέπει να σεβαστεί τον κανονισμό του Δουβλίνου από τον Ιούνιο, μας είπατε. Να σας υπενθυμίσω ότι η Ελλάδα δεν έχει κανένα κοινό σύνορο με άλλο κράτος μέλος του χώρου Σέγγεν. Ότι τα κράτη-μέλη του χώρου Σέγγεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν να κλείνουν τα εσωτερικά του σύνορα. Να συμφωνήσω λοιπόν με την άποψη του κ. Ντεπρέ και στην Ελλάδα τι θα κάνουμε. Αν δεν έχουμε αλλάξει το πρώτο άρθρο του Δουβλίνου, αν δεν με απατάει η μνήμη μου για το ποιο είναι υπεύθυνο για τους αυτούς που ε, ε, και τη χώρα εισόδου, δεν θα μπορέσουμε να ρυθμίσουμε τίποτα. Τα πάντα είναι αλληλένδετα. Εγώ δεν προσπαθώ καν να καταλάβω αυτή την ανακοίνωση. Νομίζω ότι είμαστε τελείως ε, πλάγια, δεν έχουμε καταφέρει τίποτα και εγώ κατάλαβα ότι θα υπήρχε ένα Δουβλίνο 4 για να έχουμε ένα μόνιμο μηχανισμό μετεγκατάστασης στα ευρωπαϊκά κείμενα και ξαφνικά διαπιστώνω ότι βλέποντας όμως ότι πώς λειτουργούν τα πράγματα το τελευταίο εξάμεινο κάνουμε το κεφαλιού μας. Τα κράτη-μέλη κάνουν το κεφαλιά τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθυστερεί, καθυστερεί, καθυστερεί και όσο ε, προχωράει όλα αυτά ε, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην ακουστεί η άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχουν συγκεκριμένε διατάξει όπω η Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφαλείας, γιατί ξέρουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφαλείας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει τόσε εξουσίες. Δεν ε, μα επιτρέπεται να είμαστε συνομιθέτε. αλλά τι θα μπορέσουμε να κάνουμε να δούμε στα κείμενα. Τι θα ισχύσει τώρα που ε, υπογράφει η συμφωνια Τουρκία Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού είναι οι ευρωπαϊκέ Αξίε, ε, Μα πραγματικά αναρωτιέμαι. Λυπάμαι πολύ, αλλά νομίζω ότι κάνουμε το κεφαλιού μας και ότι θα πρέπει να αντιδράσουμε όλοι από κοινού και να πούμε ότι είναι απαράδεκτη αυτή η κατάσταση. Αυτοί οι άνθρωποι που φτάνουν στα σύνορά μας είναι Σύριοι, Ιρακινοί, Αυγανοί, ε, από την Ερυθρέα, από τη Σομαλία, από το Σουδάν με ποιους υπογράφουμε συμφωνίες που δεν δημοσιοποιούνται και με τους ε, οποίους δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς κάνουμε. Υπάρχουν αντίστοιχες συμφωνίες με την TTIP προς το παρόν και πραγματικά ελπίζω να δημοσιοποιηθούν γιατί πραγματικά αναρωτιέμαι τι γράφουν αυτές οι συμφωνίες με τις χώρες του κέρατος της Αφρικής και πραγματικά ανησυχώ ιδιαίτερα. Δεν υπάρχει λόγος να εγκρίνουμε ψηφίσματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που δείχνουν ότι ανησυχούμε για την τάδη τη δίνα χώρα όταν τα κράτη-μέλη κάνουν ό,τι θέλουν αυτή τη στιγμή καταστρέφουν την ε, ίδια την ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ιδέα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Και εμείς που συναντιόμαστε με τους πολίτες καθημερινά ξέρουμε τι σημαίνει και ξέρουμε ότι υπάρχουν πολίτες παντού στην Ευρώπη που είναι διατεθειμένοι να επιδείξουν τα αλληλεγγύη. Θα πρέπει λοιπόν τα κράτη-μέλη να σταματήσουν να ακολουθούν αυτή την ιδεολογική θέση που ακολουθούν αυτή τη στιγμή. Ζήτω συγγνώμη. Ευχαριστώ. Άλλου δύο συναδέλφου έχω στον καταλογό μου, την κυρία Γκόμε και τον κύριο Μογκοριάνο. Θα ήθελα να ρωτήσω αν θέλει κάποιος άλλος το λόγο, αλλιώς θα κλείσει ο κατάλογος. κλείνει ο κατάλογος, Επόμενο. η κυρία Άννα Πολύ θέλουμε να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Τι θα πει όμως κανονικότητα, τρομοκρατία, πόλεμος και πρόσφυγες. Δυστυχώς αυτή είναι η κανονικότητα και δεν μπορούμε να σβήσουμε αυτή την ακανονικότητα. Άρα το Συμβούλιο αυτό το οποίο απεδείχθεται λειτουργεί δεν μπορεί να το εφαρμόσει πλέον. Με βάση τις νέες συνθήκες ε, το Συμβούλιο ε, επιλέγει να μην ακολουθήσει τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν μπορούμε να ε, παρουσιάσουμε κανονικό αυτό που είναι εντελώς ε, μη κανονικό και μη φυσιολογικό. Και τώρα, τους μετανάστες, τους πρόσφυγες, ό,τι και αν λένε, τους χρειαζόμαστε. Τι γίνεται λοιπόν, βλέπουμε τι κάνει ο Καναδάς, βλέπουμε τι κάνουν ε, ορισμένα μικρότερα κράτη όπως είναι η Πορτογαλία για παράδειγμα, η οποία επιλέγει απευθείας από την Ελλάδα συγκεκριμένα, όπως να το κάνουν και άλλα κράτη-μέλη, Όλα τα κράτη δε θα μπορούσαν να, να επιλέγουν τούντε άσυλο από την Τουρκία χωρί να το κάνουν όμως και κάνουν το αντίθετο κιόλα. Ποιο είναι το αντίθετο. Είναι η απόφαση του Συμβουλίου τη προηγούμενης εβδομάδα. που είναι ονειδο, Εγώ ντρέπομαι ως Ευρωπαία. Γιατί και εγώ πιστεύω ότι καταστρέφουν την Ευρώπη και σίγουρα καταστρέφουν την αξιοπιστία της Ευρώπης και την, το ηθικό μας ε, ανάστημα. Και πολύ σωστά τα λέμε αυτά. Είναι πραγματικά ε, επονίδιστο αυτό που κάνει το Συμβούλιο και αυτό που κάνει η Κομισιόν και στρέφουμε στην Κομισιόν γιατί εμείς περιμέναμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δράσει και να πει στο Συμβούλιο ελάτε στα συγκαλά σας και δεν το κάνει. Και ο Κάρλος Κοέλιο το είπε και εμεί, Ναι, είμαστε υπέρ του Σέγγεν. Βλέπουμε όμω ότι αυτοί οι οποίοι καταστρέφουν το Σέγγεν και που εξωστρακίζουν την Ελλάδα, δεν το τραβάει κανείς ταυτί από την Κομισιόν. Και πού έχουμε φτάσει. Έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση σήμερα, όπου το Συμβούλιο τελικά και οι πρωθυπουργοί τιτιβίζουν και του τουιτάρουν οι Σύροι θα επιστραφούν από σήμερα στην Τουρκία. Sorry, μήπως δεν γίνεται πόλεμος πια στη Συρία και δεν το κατάλαβα. Δεν υπάρχει εξαφλίως καταστροφή, τρομοκρατία στη Συρία πια. Και δεν είναι αυτοί καλοί λόγοι για οποιονδήποτε που έρχεται από τη Συρία για να του χορηγηθεί καθεστώς πρόσφυγα. Και τους γυρίζουμε πίσω, σαν να άλλαξε κάτι στις συνθήκες που τους κάνουν θεμητούς ετούντες άσυλο αυτούς τους ανθρώπους από τη Συρία. Εντάξει. Δεν είναι η Τουρκία το θέμα και ούτε καν μιλάω για την Τουρκία. Εγώ μιλάω για μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πού βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση της αλληλεγγύης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σέβεται την Οικουμενική Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Προσφύγων και Μεταναστών κτλ όχι απλά είναι ανήθικο, όχι απλά είναι παράνομο, αναξιοπρεπές, αλλά και ανέφικτο στην πράξη είναι όλο αυτό το σύστημα. Για μήνες είχαμε συνεντεύξεις για μετεγκατάσταση 160.000 ανθρώπων, κάτι που είχε συμφωνηθεί στο Συμβουλίο και δεν λειτουργήσε. Και μου λέτε τώρα ότι θα βιαστούν για να επιστραφούν στην Τουρκία όλοι αυτοί που πρέπει να επιστραφούν στην Τουρκία. Αυτό είναι γελίο. Είδαμε χθε κάτι εικόνες από ανθρώπους οι οποίοι πεθαίνουν στις ακτές τις ελληνικές και πραγματικά αυτό είναι μια καταγγελία, ε, είναι καταδίκη για τους ηγέτες μας. Εγώ λέω ότι πρέπει να προσφύγουμε στο δικαστήριο κατά το Συμβουλίο. Ενδιαφέρον θα ήταν αυτό το βήμα, λέει η Πρόεδρος, να πάμε στο δικαστήριο το Συμβούλιο. Ο κύριος Σουγκαριάνο, τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ για να κάνω κι εγώ φασαρία και αν τα κάνω πιο δύσκολα τα πράγματα. Άκουσα τον τελευταίο μιλητή, ή την τελευταία μιλήτρα που μίλησε για αλληλεγγύη. Πράγματι, αν μιλάμε για αλληλεγγύη, να σας υπενθυμίσω ότι η Ρουμανία και η Βουλγαρία έμειναν εκτός του Σέγγεν επανειλημμένος και όχι μόνο μια φορά παρόλα αυτά ε, έχει δηλωθεί ότι είναι σε θέση να ε, ενταχθούν. Δεν μπορούν να πάρουν πρόσφυγες και δεν μπορούν να προστατεύσουν τα εξωτερικά σύνορα. Αν υποθέσουμε ότι αύριο έχουμε κύματα προσφύγων στην, ε, στα σύνορα με το, στον Πόντο και στη Μαύρη Θάλασσα, Ρουμανία-Βουλγαρία. αφού συνεχώς τους αρνούνται το καθεστώς ε, της χώρας Σέγγεν. Τι θα κάνουν αυτές οι χώρες. Λέμε αυτό δεν υπάρχει, αλλά νομίζω θα ήταν τεράστια χάρη Από εντό αγωγικών δευτέρας κατηγορία κράτη-μέλη, όπως είναι η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Πρόεδρος, χαίρομαι πολύ, χαίρομαι πολύ, γιατί σήμερα είχα τη δυνατότητα να δώσω το λόγο σε όλους τους συναδέλφους και για όση ώρα ήθελαν. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση. Σίγουρα είναι συναισθηματικά φορτισμένη και καταλαβαίνω ότι προς το παρόν τουλάχιστον ο κίνδυνος δεν λέω ότι θα συμβεί, αλλά ο κίνδυνο τη διατρέχει Ευρώπη είναι να χάσει την καλή εικόνα που έχει στον υπόλοιπο κόσμο, εστιάζοντα μόνο σε μια ή δύο Συμφωνώ με τον συνάδελφό μα, τον κύριο Κοέλιο, που λέει ότι δύο χρόνια ελέγχου των συνόρων ίσως είναι λίγο υπερβολικό. Όχι μόνο γιατί είναι αφισβητήσιμη νομική βάση, θα επανέλθει σίγουρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό, όμως οι ε, πολίτες μας τι θα σκεφτούν ε, με αυτό το κλείσιμο των συνόρων για δύο χρόνια. Πώς ζούμε, πώς ε, συνεργαζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έρχομαι στα 850.000 850.000 πρόσφυγες που έρχονται στην Ευρώπη μέσω της Ελλάδας. Σας φανταστούμε με το σύστημα του Δουβλίνου που μέχρι πέρυσι ας πούμε λειτουργούσε τέλεια. Όλοι οι μετανάστες καταγράφονταν στην Ελλάδα, όλες οι αιτήσει ελέγχονταν. Ξεκινούσε στην Ελλάδα η δικασία ε, για την εκπαίδευση των αιτήσεων ασύλου και στην Ελλάδα παρέμεναν όλοι οι πρόσφυγες που θα γίνονταν αποδεκτοί ως πρόσφυγες, έντοντες άσυλο. Ας συγκρίνουμε τώρα αυτή την κατάσταση με την κατάσταση στη Γερμανία, τη χώρα την οποία κατάγομαι. Η μεγάλη και η πλούσια Γερμανία προς το παρόν δεν είναι έτοιμη εντελώ για να καταγράψει όλους τους ερχόμενους μετανάστες. Δεν είμαστε έτοιμοι εντελώς ακόμη για να κινήσουμε διαδικασίες εξέτασης αιτήσεων ασύλου βραχυπρόθεσμα, αλλά ζητάμε να το κάνει η Ελλάδα παρόλα αυτά και αναφερόμαστε στο σύστημα δουλειών πώς ισχύει τώρα. Όλοι οι πρόσφυγες θα πρέπει να παραμείνουν τέσσερα χρόνια στην Ελλάδα. Και όταν χρειάζεται να αποσταλούν πίσω κάποιοι, ε, και αν τους δεχτούν βέβαια, ε, οι χώρες τους, αυτό θα πρέπει να το αναλάβει η Ελλάδα. Αυτό είναι το μέλλον αυτής της χώρας. Επομένως, το ερώτημα του να κλείσουν ή το να γίνονται έλεγχοι ε, στα σύνορα, στον χώρο Σέγγεν, ε, ο έλεγχος των εσωτερικών σύνορων θα έχει ως αποτέλεσμα δεν ξέρω, μήπω έχω παραβλέψει κάποια άλλα σημεία που μπορεί να μου απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ένα ή δύο-τρία, ας πούμε, ε, κράτη της Ένωσης με εξωτερικά σύνορα θα πρέπει να αντιμετωπίσουν και να φέρουν όλα τα βάρη, ενώ οι άλλοι θα καθίσουν στα βρωμένα χέρια λέγοντας δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα. Ορίστε, αυτό είναι το Δουβλίνο, αυτά τα προβλέπει το Δουβλίνο. Εμείς ψάχνουμε εσωτερικές λύσεις, αλλά αν αποφασίσουμε μόνο αυτό το δρόμο με το Σέγγεν και δεν βρούμε λύσεις μεταγκατάστασης ή μεταφοράς σε κάποια άλλη χώρα, και αν δεν φροντίσουμε να εξασφαλιστούν καλές συνθήκες διαβίωσης για αυτούς τους πρόσφυγες, τότε ίσως η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μεγάλα προβλήματα στο τέλος. Προσπαθώ να καθησυχάσω κάπως ε, τα έντονα αισθήματα που ακούσαμε να εκφράσουν ορισμένοι συνάδελφοι. Θα δώσω τώρα το λόγο καταρχάς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελπίζοντας να απαντήσει στα περισσότερα ή σε όλα στην ε, δυναμική περίπτωση ερωτήματα των μάλλον. Κύριε Μουσέλ, έχετε το λόγο. Thank you, Madam Chair. First of... Ευχαριστώ, Πρόεδρο, και χαίρομαι ιδιαίτερα, καταρχάς που βλέπω ότι τόσοι βουλευτές ε, εξακολουθούν να συμφωνούν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρέπει να επανέλθουμε σε ένα κανονικό Σέγγεν. Το κανονικό Σέγγεν όμω δεν είναι κάτι το οποίο το πετυχαίνουμε έτσι με, ένα, μια ωραία δήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χρειαζόμαστε και τα κράτη-μέλη να συμφωνήσουν και αυτό δεν είναι εύκολο, ξέρετε. Όλοι μαζί θα πρέπει να συνεργαστούμε για να πετύχουμε μια επαναφορά στο Σέγγεν. Ιδάλω θα ξεψυχήσει το Σέγγεν. Γιατί αν δεν βρούμε μία λύση και λέμε απλά ας επανέλθουμε σε μια κανονική κατάσταση, θα δείτε τι θα συμβεί, θα δείτε τι θα γίνει τώρα να επικεντρήσει το δίκαιο του εξτρεμισμού. Θα πρέπει να φροντίσουμε λοιπόν το Σέγγεν να ξαναμπεί υπό σωστού όρου. Και όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει να μεταρρυθμίσουμε το Δουβλίνο. Όλοι συμφωνούμε ότι δεν είναι δίκαιο για την Ελλάδα να αντιμετωπίσει όλες τις αιτήσει ασύλου. Αλλά θα πρέπει να βρούμε και ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο για να μεταρρυθμίσουμε το Συμβούλιο. Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται σκληρά για να προσπαθήσει να βρει τους σωστούς όρους για τη μεταρρύθμιση, την αθεώρηση του Δουβλίνου. Και αυτό με οδηγεί στο ερώτημα που έθεσε ο κ. Ντεπρέ. Ναι, προτείναμε να υπάρξει η ανακοίνωση της Επιτροπής για το μέλλον του Δουβλίνου, για το μέλλον του ασύλου στις 16 Μαρτίου, αλλά αποφασίσαμε να αναβάλουμε μέχρι τις 6 Απριλίου. Γιατί έγινε έκτακτη σύνοδος την ακριβώς επόμενη ημέρα. Δεν υπήρχε νόημα λοιπόν, δεν είχε νόημα την προηγούμενη ημέρα να κατεθεί στο τραπέζι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στα μέσα της διαπραγμάτευσης ε, της Τουρκίας ε, την μεταρρύθμιση του Δουβλίνου, θα έχει χαλάσει τη συζήτηση αυτή και είμαστε από... υποστηρίζουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί το Δουβλίνο τη σωστή χρονική στιγμή. Άρα αναβάλαμε για λίγε εβδομάδε την κατάθεση τη πρόταση, η οποία και θα γίνει πλέον τον Απρίλιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι το τρέχον σύστημα έχει καταργηθεί και δεν ισχύει. Το γεγονό ότι έκανε μια ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν σημαίνει ότι άλλαξε νομοθεσία εξακολουθεί να επικρατεί η νομοθεσία. Θα αλλάξει μόνο εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Συνομοθέτης αποφασίσουν για ένα νέο σύστημα Δουβλίνου. Μέχρι να συμβεί αυτό, το σύστημα που έχει εγκριθεί και οι τρέχοντες κανόνες συνεχίζουν να ισχύουν. Και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η Ελλάδα θα ξαναμπεί στο σύστημα αυτό. Και γιατί. Γιατί έχει ανασταλεί το Δουβλίνο για την Ελλάδα, όχι μόνο λόγω του μεγέθους, όχι μόνο επειδή θα ήταν αυτό ένα άδικο φορτίο για την Ελλάδα, αλλά επειδή οι όροι υποδοχής ε, και οι διαδικασίες ασύλου δεν ήταν αυτοί που έπρεπε, δεν ήταν το επίπεδο που θα έπρεπε. Τι θέλουμε λοιπόν, θέλουμε οι μετανάστες να φτάνουν στην Ελλάδα να έχουν κάποια αξιοπρεπή διαδικασία και να υπάρχουν ε, σωστές διαδικασίες. Έχει κάνει μεγάλη πρόοδο η Ελλάδα από αυτή την άποψη. Και πραγματικά το πετυχαίνει αυτό σιγά σιγά. Γι' αυτό θέλουμε να θεωρήσουμε ότι η Ελλάδα επανέρχεται στο σύστημα του Δουβλίνου. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ξαναστείλουμε τους, ε, τον εκατομμύριο πρόσφυγες ε, πάλι στην Ελλάδα που ήλθαν πέρσι, όχι. Αλλά στο μέλλον θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να ξαναστέλνουμε τον κόσμο στην Ελλάδα για να αποτρέψουμε και την δεύτερογενή κίνηση. Γιατί αν ο κόσμος ξέρει ότι μπορεί να επιλέξει τη χώρα στην οποία θα πάει και να ταξιδέψει όπως θέλει στην Ελλάδα, θα το κάνει. Αν ξέρει ότι θα επιστραφεί η βάση του Δουβλίνου, αυτό θα αποτελέσει μεγάλο, μεγάλη πηγή μείωση στον δευτερευουσών αυτών μετακινήσεων σε ό,τι αφορά την επανεγκατάσταση. Ας το δούμε, ας δούμε την αλήθεια κατάματα. Η επανεγκατάσταση δεν λειτουργούσε γιατί στον, στην οδό του Δυτικού Βαλκανίων ε, ήταν ανοιχτά τα σύνορα. Αν είστε τέσσερις πατέρας με γυναίκα και παιδιά. Και μπορείτε σχετικά εύκολα να μην ξέρετε μάλλον πού θα πάτε. Ή Έχετε την δυνατότητα να πάτε στη Γερμανία και να ξέρετε ότι θα πάτε στη Γερμανία σε λίγες ημέρες, αλλά θα πάτε στη Γερμανία. Τώρα, που είναι πιο δύσκολο να φτάσει κανεί στη Γερμανία, έχει ξεκινήσει η επανεγκατάσταση. 300, 300 μεταγκαταστάσεις ανά ημέρα γίνονται πλέον. Γιατί ο κόσμο ξέρει ότι αυτή είναι η καλύτερη εναλλακτική που έχει στη διάθεσή του. Αν θέλουμε λοιπόν να λειτουργήσει η επανεγκατάσταση, θα πρέπει να υπάρχουν συνοριακές συνοριακέ ε, διαδικασίες. Και αυτό ήταν και αυτό ήταν ο σκοπός της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε ό,τι αφορά τη συμφωνία με την Τουρκία. Άκουσα και την κυρία Γκόμες και τους υπόλοιπους συμβουλευτές ε, Πετύχαμε μια συμφωνία στο Συμβούλιο και η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου θεωρεί ότι είναι νόμιμο και την Τουρκία μπορεί να θεωρηθεί ως ασφαλή χώρα για τους σκοπούς αυτούς. Έγινε μία σχετική διακήρυξη στο Συμβούλιο στις 19 Μαρτίου που δεν είναι αντίθετη προς αυτό που αναφέρει ότι αν πληρούνται οι όροι, αν η Τουρκία πληρεί μία σειρά όρων σε ό,τι αφορά ε, τη συνθήκη της Γενέβης και την αρχή της μη επαναπροώθησης είναι ασφαλής χώρα. Έχουμε λοιπόν τώρα χώρες που συνεργάζονται και με την Ελλάδα και με την Τουρκία. Έχουμε μια ομάδα νομικών που έχει μεταβεί εκεί προκειμένου να υπάρχει ένα ασφαλές νομικό σύστημα και να πληρούνται και άλλοι όροι προκειμένου όταν επιστρέφονται οι μετανάστες να γίνονται βάσει των όρων της συνθήκης της Γενέβης και των διεθνών κανόνων. Κυρία Γκόμες, μιλάμε για όσους πηγαίνουν και πάνε, επιστρέφονται στην Τουρκία. Όχι για μετανάστες και πρόσφυγες που επιστρέφονται στη Συρία. Το τονίζω αυτό. Θεωρούμε ότι η Τουρκία είναι ασφαλή τρίτη χώρα. Ότι όποιο άτομο θα φτάνει στα ελληνικά νησιά θα έχει δικαίωμα να ζητάει άσυλο και θα περνάει από μεμονωμένη αξιολόγηση. Εξακολουθεί να υπάρχει μεμονωμένη και ατομική εξέταση. Αν θεωρηθεί ότι είναι επικίνδυνο να επιστραφεί το άτομο αυτό στην Τουρκία, δεν θα επιστραφεί στην Τουρκία. Και έχουμε και ένα σύστημα ε, δικαστών και υπάρχει δυνατότητα έφεσης κτλ. Για να υπάρχει νομική βεβαιότητα. σε ό,τι αφορά δηλαδή τα όσα προβλέπει το άρθρο 38, το οποίο και από σύγχρονη με αποφαση από το Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο. Εφαρμόζουμε αυτά που προβλέπονται στην οδηγία για την χορήγηση ασύλου. Σε ό,τι αφορά τα σχόλια της κυρίας Βερζιά για τους ε, νόμιμους τρόπους. Συμφωνούμε απόλυτα, χρειαζόμαστε πιο πολλούς νόμιμους τρόπους και σε ανακοίνωση της 6 ε, Απριλίου που θα εγκριθεί στις 6 Απριλίου, τονίζουμε αυτές τις νόμιμες οδούς και σε ό,τι αφορά τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας της προηγούμενης Παρασκευής, να σας πω ότι εκεί μιλάμε για επαναγκατάσταση και περισσότερες ε, Ε, αναφέρουμε αριθμητικά 18.000 σε μετριότητα προσθήκης 54.000. Νομίζω ότι είναι μεγάλο επιτεύγμα αυτό σε ό,τι αφορά σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε μελών. Αυξάνουμε λοιπόν τους νόμιμους τρόπους. Ξέρω ότι είναι μια αρχή, αλλά θα πρέπει να καλωσορίσουμε και αυτήν την θετική εξέλιξη. Σας ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συμφωνώ. Καταρχάς, ό,τι και να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χρειαζόμαστε και τα κράτη-μέλη. Δεύτερον, δεν είμαι απόλυτα βέβαιη ότι μόνο ο αριθμός των προσφύγων ε, είναι αυτός ο οποίος οδήγησε στην αύξηση των ε, προβλημάτων στην Ευρώπη. Πρέπει να το λάβουμε και αυτό υπόψη. Τρίτον, συμφωνώ ότι πρόκειται για ένα πρώτο βήμα. Όντως, ό,τι κάνουμε στον τομέα των προσφύγων και των μεταναστών είναι ένα πρώτο βήμα, δεν είναι το σύνολο της εικόνας. Και συμφωνώ τους ότι ίσως εάν μπορέσουμε να στείλουμε ε, πίσω τους πρόσφυγες στην Ελλάδα αλλά μετά υπάρχει ένα καλό πρόγραμμα ε, επανεγκατάστασης και μετεγκατάστασης ίσως θα ήταν χρήσιμο. Ίσως τα κράτη-μέλη όμως θα μπορούσαν να μας πούνε δεν είναι απλώς ωραία πράγματα σε χαρτί όλα αυτά, αλλά είναι όντως διατεθειμένοι να εργαστούν για μετεγκατάσταση και επανεγκατάσταση, εάν μπορέσουμε να έχουμε και τις κατάλληλες προϋποθέσεις, διότι αυτό αποτελεί προϋπόθεση ώστε να βρούμε τελικά μια καλή λύση. Με αυτό θα ήθελα να δώσω το λόγο στην, στο Συμβούλιο, αν θέλουν να σχολιάσουν και αυτοί για τις ερωτήσεις και παρατηρήσεις που ακούσαμε από τους συναδέλφους. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς να υπενθυμίσω αυτό που είπατε και στο πρώτο σας συμπέρασμα. Πράγματι το ε, Συμβούλιο θέλει και αυτό να επιστρέψει στην ομαλότητα και ε, επ' αυτού εργάζεται. Ασχολούμαστε με διάφορα θέματα, το είπατε και εσείς και στα συμπεράσματά σας. Ε, το Συμβούλιο επεξεργάζεται νομοθετικές προτάσεις που έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, υπάρχει πρόταση για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. Περιμένουμε την ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για το Δουβλίνο και θα το συζητήσουμε και αυτό κατά προτεραιότητα. Και όσον αφορά τη συμφωνία που επετεύχθη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την περασμένη εβδομάδα, νομίζω ότι θα πρέπει να συμφωνήσω με αυτό που είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πράγματι, και εγώ περιμένω ότι τις επόμενες εβδομάδες θα υπάρξει βελτίωση στην περίπτωση της μετεγκατάστασης. Ευχαριστώ. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Ξέχασα να σας υπενθυμίσω ότι Όλοι αυτοί οι οποίοι ζητούν να αποσταλούν οι πρόσφυγες πίσω στη Συρία σχετίζονται με δηλώσεις κάποιων Τούρκων εκπροσώπων που είναι, ε, είπαν ότι είναι διατεθειμένοι να εκτίσουν ασφαλείς περιοχές για τους πρόσφυγες στη Συρία και κάποιοι μιλούν για επαναπρόθεσή τους, ότι επιστρέφουν στην ε, Τουρκία μεν, αλλά υπάρχουν κάποιες εκθέσεις που δημιουργούν κάποιες αμφιβολίες επί της, ε, του θέματος. Επειδή έχουμε λίγα λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας, ε, είδα ότι η κυρία Βερζιά ήθελε να κάνει μια επιπλέον ερώτηση. Δεν ξέρω αν θέλει και πάλι το λόγο. Κυρία Βερζιά... Ναι, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι είμαι ικανοποιημένη διότι πλέον έχουμε έναν αριθμό ε, ε Ε, μερικών χιλιάδων ανθρώπων. Ξέρουμε όμως ότι είναι πολύ πιο κάτω από τις απαιτήσει. Ακόμα και μειωμένος ο αριθμός των ατόμων που φτάνουν στην Ελλάδα είναι χίλιοι με τρεις χιλιάδες καθημερινά και νομίζω ότι αυτές οι κινήσεις δεν θα σταματήσουν. Πώς ε, σκοπεύει να σταθεί στο ύψος των αναγκών αυτών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πώς ε, πραγματικά θα σεβαστεί το διεθνές δίκαιο. Αλλιώς να μας εξηγήσουν ε, αν η Τουρκία είναι ασφαλής χώρας ή θα είναι ασφαλής χώρας και σε, γιατί σέβονται τους κανόνες. Ποια είναι τα κριτήρια βάσει των οποίων ε, η Τουρκία είναι ασφαλής χώρας. Γιατί από όλα τα σχόλια που έχω από την Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν είναι προς αυτή την κατάσταση. Πραγματικά λοιπόν θα θέλαμε να έχουμε αυτά τα κριτήρια που αναφέρατε ώστε να μπορέσουμε να κρίνουμε κι εμείς ε, πολύ γρήγορα. Να επανέλθουμε, κύριο Δεπρέ θέλει το λόγο. Ναι, κυρία Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος. Απλά θέλω να βεβαιωθώ ότι κατάλαβα τύπη κομισιόν. Στο έγγραφό, της λέτε, στο έγγραφό της λέει ότι τον Ιούνιο του 2016 θα μας παρουσιάσει την αξιολόγηση για επανάληψη των μεταφορών προς την Ελλάδα δυνάμει του κανονισμού του, του Δουβλίνου. Δεν έχει αναδρομική ισχύ αυτό, άρα μόνο για ό,τι έχει συμβεί μετά από κάποια ημερομηνία. Δεν ξέρω, 20 Μαρτίου και μετά, δεν ξέρω ποια, ποια ημερομηνία μιλάμε. Είναι σαφές αυτό, άρα δεν ισχύει αναδρομικά. Ευχαριστώ. I'm Θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσθέσει κάτι. Εγώ νομίζω ότι το ερώτημα κατά πόσον η Τουρκία είναι ασφαλής τρίτη χώρα ή ασφαλής ε, χώρα προέλευσης Υπάρχουν κριτήρια, πρέπει να το ελέγξουμε. Νομίζω όμως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε, δεν με ικανοποίησε όμως απόλυτα αυτή η απάντηση, είπε πάντως ότι σε σχέση με το προσφυγικό είναι σαφές ότι η Τουρκία πρέπει να επεξεργαστεί τον κατάλογο για το ποιος είναι τον άσυλο, πρέπει να επεξεργαστεί τα κριτήρια ε, της Σύμβασης ε, της Γενέβης ε, για το σύστημα θεωρήσεων που κανείς δεν το ανέφερε σήμερα για την Ελευθέρωση των θεωρήσεων, νομίζω υπάρχουν 75 σημεία που πρέπει η Τουρκία να εκπληρώνει. Μέχρι τη στιγμή εκπληρώνει τα 32, άρα έχει πολλή δουλειά μπροστά της. Συμφωνώ τώρα ότι πολλή δουλειά έχουμε και εμείς σε επίπεδο κρατών μελών. Καταλαβαίνω τις ανησυχίες σας. 300 πρόσφυγες μετεγκαθίστανται ε, μέσα σε μια μέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ίσως πολύ λίγος αυτός ο αριθμός, αλλά από τον περσινό Σεπτέμβριο μετεγκαταστάθηκαν ίσως 900 πρόσφυγες. Τώρα να έχουμε 300 την, ημέρα, ημέρα είναι πρόοδος. Δεν αρκεί, αλλά είναι πρόοδος. Υπάρχει κάποια αλλαγή, κάποια κίνηση. Ίσως χρειάζεται περισσότερος χρόνος. Απάντησε το Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλει να επανέλθει. Να σας ευχαριστήσω όλους και όλες και όλα τα θεσμικά όργανα που πήραν μέρος σε αυτή την πολύ σημαντική συζήτηση και με μία παρατήρηση θα ολοκληρώσω. Ο έλεγχος όλων των μέτρων που εφαρμόζονται ή που προβλέπονται από το Συμβούλιο είναι πολύ σημαντικό να γίνεται με αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν έχουμε κάνει οδηγίες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ελέγχει λοιπόν θέλουμε να τηρούνται οι αξίες μας, να γίνονται σεβαστές, αλλά τέλος πάντων αυτό ίσως θα πρέπει να το συζητήσουμε και να το απαντήσουμε σε ένα άλλο πλαίσιο. Ευχαριστώ λοιπόν από τη συνάδελφη ολοκληρώνουμε αυτό το σημείο τη ημερήσια διάταξης και περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο τη ημερήσια διάταξης. Το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης σε κάποιο βαθμό σχετίζεται με το χώρο Σέγγεν, νομική βάση του συστήματος πληροφοριών Σέγγεν δεύτερης γενιάς που προβλέπει τη δυνατότητα χρήση αγγλικών αποτυπωμάτων τα οποία ε, βρίσκονται σε μια βάση δεδομένων για την ταυτοποίηση των προσώπων. Πολύπλοκο από τεχνική πλευρά το θέμα, διότι θα πρέπει να ελέγχονται όλα τα λήματα και όλα τα δακτυλικά αποτυπώματα της βάσης δεδομένων. όταν συμφωνήθηκε η νέα νομική βάση, υπήρξε μια συμβαστική πρόταση. Δηλαδή, η λειτουργική αυτή δυνατότητα ενεργοποιείται μόνο εφόσον υπάρχει διαθέσιμη σχετική τεχνολογία. Και φαντάζομαι ότι αυτό ήταν προφανέ αλλά τέλο πάντων. Για το σκοπό αυτό και δυνάμει το άρθρο 22 εδάφιο C τη απόφαση για το σύστημα C Δεύτερη Γενιά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε να παρουσιάσει μια έκθεση για την διαθεσιμότητα και ετοιμότητα τη απαιτούμενη τεχνολογία και θα πρέπει να ζητηθεί γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτό το θέμα. Οι συντονιστέ τη Επιτροπή ΛΥΜΠΑ αποφάσισαν να καταθέσουν, να προετοιμάσουν μάλλον ένα ψήφισμα στο οποίο θα αναφέρεται η άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα δώσω το λόγο για μια ακόμη φορά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας παρουσιάσει αυτή την έκθεση και έπειτα θα λάβουν το λόγο οι συνάδελφοι να θέσουν τα ερωτήματά τους. Ο κύριος νομίζω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πάρει τώρα το λόγο. Η κυρία, συγγνώμη. Κυρία Γιάννη, παρακαλώ έχετε το λόγο. Καλησπέρα αγαπητοί συνάδελφοι από την Επιτροπή ΛΥΠΕ. Είμαι η κυρία Γιάννη, επικεφαλής ε, και υπεύθυνη για το σύστημα πληροφοριών Σέγγεν. Είμαι από την μονάδα B3 της DigiHome για τα συστήματα πληροφόρησης για την ασφάλεια και είμαι εδώ για να μοιραστώ κάτι θετικό, μια θετική είδηση μαζί σας μετά από την προηγούμενη συζήτηση. Επιτυχής λειτουργία του συστήματος πληροφοριών Σέγγεν δεύτερης γενιάς. Το σύστημα ε, ξεκίνησε να δουλεύει σε 9 Απριλίου του 2013 και έκτοτε έχει αναπτυχθεί και αποτελεί το βασικό σύστημα ασφαλείας της Ευρώπης για την ε, ασφάλεια, την εφαρμογή του νόμου και τη συνοριακή ασφάλεια. Όλα αυτά είναι πραγματικά αδιανόητα χωρίς το σύστημα πληροφοριών ΣΕΝ. Το 2013 λοιπόν τα ξεκίνησε το σύστημα, περιλαμβάνει 47 εκατομμύρια καταγραφές, τώρα είμαστε στις 65.000. 65 εκατομμύρια, συγγνώμη, με 28 κράτη-μέλη ξεκινήσαμε. Τώρα έχουμε και το Ηνωμένο Βασίλειο, 29 λοιπόν μέλη που συμμετέχουν στο σύστημα και συνδέονται λοιπόν η αστυνομία, οι δικαστές και το καθεξής. Το σύστημα άλλαξε, είχε χρησιμοποιηθεί 3 δισεκατομμύρια φορές το 2015. Για να σας δώσω συγκριτικά μια μια τάξη μεγέθους, το 2014 ήταν 2 δισεκατομμύρια η χρήση του συστήματος, 1 δισεκατομμύρια δηλαδή. Άλλο ένα στατιστικό στοιχείο για την χρήση του συστήματος το 2015, πάνω από 150.000 αστυνομικές δράσεις ε, κινήθηκαν βάσει πληροφοριών του συστήματος πληροφόρησης εγγενική καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Επίσης, ε, χρησιμοποίησε το σύστημα. Πρόκειται σχεδόν για το μόνο σύστημα όπου οι εθνικέ αρχέ συνεργάζονται και αυτό αναγνωρίζεται και από το συντονιστή για θέματα τρομοκρατία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν το ότι υπάρχει καν το σύστημα αυτό και είναι απόλυτα απαραίτητο να αξιοποιείται στο έπακρον. Όπω υπέδειξε και η κυρία Πρόεδρο, άλλωστε βάσει του άρθρα 22 σημείο C γαμα των δύο νομικών αυτών μέσων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποχρεούταν να παρουσιάσει μια έκθεση για την διαθέσιμότητα και την ετοιμότητα της τεχνολογίας για την αναζήτηση βάση δακτυλικών αποτυπωμάτων από τότε που ξεκίνησε το σύστημα. Αυτή ήταν η βασική αν θέλετε, εξέλιξη σε ό,τι αφορά την ενημέρωση του συστήματος ε, θα πρέπει να γίνει για την έκθεση αυτή μια διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και χαίρομαι για την ευκαιρία που έχουμε να σας ε, περιγράψω σήμερα πόσο επιτυχές είναι το σύστημα και πόσο καλά λειτουργεί. Να σας δώσω λίγο και το ιστορικό υπόβαθρο. Υπάρχουν ήδη συστήματα καταχώρησης των αποτυπωμάτων στο σύστημα πάνω από 83.000 πλέον ε, στο σύστημα υπάρχουν 83.000 δηλαδή καταχωρήσεις δακτυλικών αποτιμάτων, μόνο όμως μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα. Ένα άτομα λοιπόν εντοπίζεται βάσει ονόματος και ημερομηνία γέννησης και αυτή η αναζήτηση μπορεί να επιβεβαιωθεί από το δακτυλικό αποτύπωμα στο σύστημα. Αυτό που θέλουμε πλέον είναι να υπάρχει ένα βήμα παραπάνω. Να υπάρχει και ταυτοποίηση των ατόμων αυτό που αποκαλείται ως one too many search στο σύστημα. Η λειτουργία με τα δακτυλικά αποτυπώματα που αποτέλεσε και μία βασική αλλαγή και βελτίωση στο σύστημα δεύτερης γενιάς χρησιμοποιείται ουσιαστικά και από τις 29 χώρες, δύο χώρες δεν το χρησιμοποιούν επί του παρόντος Αλλά τώρα θέλουμε, αλλά ως τώρα, όπως σας είπα, το θέμα είναι η επιβεβαίωση της ταυτότητας. Μόνο αυτό προβλέπετε. Πιστεύουμε ότι αυτό το περαιτέρω σύστημα για τη χρήση του συστήματος για σκοπούς ταυτοποίησης θα καλύψει ένα κοινό στην Ευρώπη. Γιατί ε, προς το παρόν δεν υπάρχει ευρωπαϊκό σύστημα αυτοματοποιημένης αναγνώρισης τελικών αποτυπωμάτων για λόγους ασφάλειας. Θα δούμε λοιπόν όταν θα συζητήσουμε το θέμα τη ελέγχου ασφαλείας των μεταναστών ότι υπάρχουν τέτοια κενά στην Ευρώπη. Και πολλοί α, μετανάστες που δεν έχουν καταχωριστεί ή των οποίων η ταυτότητα είναι αφιλεγόμενη δεν μπορούν να αναγνωριστούν οριστικά γιατί δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά τέτοια συστήματα και μια και το Eurodact είναι βάση δεδομένων για τους μετανάστες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για περιορισμένους σκοπούς ε, σε ό,τι αφορά την επιβολή του δικαίου. Και επίσης αυτό αυξάνει το πεδίο, το περιθώριο ε, δράσης των εγκληματιών, γιατί μπορούν να χρησιμοποιούν πλαστά έγγραφα. 25% των ε, ειδοποιήσεων στο συστήματα στο σύστημα Schengen, τον alerts, ε, έχουν ε, παράλληλες ταυτότητες, χρησιμοποιούν και πλαστές ταυτότητες. Γι' αυτό είναι σημαντικό να υπάρχει αυτή η λειτουργία προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι με τα δακτυλικά αποτυπώματα θα ε, εντοπίζεται το κάθε άτομο στα σύνορα, ακόμα και αν χρησιμοποιούν άλλο όνομα άλλη ταυτότητα. Και να επανέλθω τώρα στην έκθεση που αποτελεί και το αντικείμενο της συζήτηση για να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει πραγματικά διαθέσιμη η τεχνολογία. Το 2004 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέθεσε στο κοινό ερευνητικό κέντρο, το οποίο αποτελεί επίσης η Γενική Διευθύνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να προτιμάσει μια μελέτη η οποία και θα εξέταζε όντως πώς μπορεί να λειτουργήσει και πώς εφαρμόστηκε για σκοπούς ταυτοποίησης αυτό το σύστημα δακτυλικών αποτυπωμάτων και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Προετοιμάστηκε λοιπόν μια εκτενέστατη έκθεση η οποία είναι δημόσια διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Κοινού Ερευνητικού Κέντρου. Κοιτάξτε την αν σας ενδιαφέρουν τα στοιχεία αυτά. Και βάσει λοιπόν της έκταση αυτής, της μελέτης αυτής, της έρευνας αυτής, προετοιμάζουμε και τι συστάσει. Ε, του κοινού ερευνητικού κέντρου, το οποίο και εξέτασε τα δύο βασικά ε, συστήματα τα ευρωπαϊκά, το Eurodac και το VIS, το οποίο βασίζεται ήδη στην τεχνολογία αυτή και, και το VIS ως τώρα έχει πάνω από 70 εκατομμύρια αποτυπώματα και στο Eurodac έχουμε 4,3 εκατομμύρια δακτυλικά αποτυπώματα. Πέραν από αυτό, το ερευνητικό κέντρο εξέτασε το σύστημα των εθνικών τεχνολογιών και στο τέλος της έρευνας απέταξε ότι υφίσταται αυτή η τεχνολογία, διατίθεται και χρησιμοποιείται σε ευρύτατη κλίμακα, πολύ ευρύτερη από ότι θα ήταν αν χρησιμοποιούνταν στο πλαίσιο του ΣΥΣ στο σύστημα πληροφοριών Σέγγεν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη λειτουργία ταυτοποίησης. Στην, ε, στην παρούσα φάση υπάρχουν μόνο 8.000 καταχωρήσεις τέτοιων ατόμων και τα δακτυλικά αποτυπώματα θα μπορούσαν να ε, ταιριάξουν μόνο σε αυτά τα 8.000, αυτές τις 8.000 καταχωρήσεις. Δεν αναμένουμε να αυξηθεί δραματικά αυτός ο αριθμός ε, των ε, καταχωρισμένων ατόμων. Είναι σταθερό τα τελευταία χρόνια. Και επίσης θα συνδεθούν τα δακτυλικά αποτυπώματα με τη σύλληψη που είναι που είναι, μας ενδιαφέρει πιο πολύ και στις ειδοποίησει για άρνηση εισόδου για να αποφευχθεί η εκ νέου είσοδος ε, υπηκόντρωτων χωρών σε άτομα, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες τους έχουν ήδη απορρίψει. Θεωρούμε ότι ε, βάσει των στοιχείων αυτών το ΣΥΣ αυτό δεύτερης γενιάς θα ήταν πολύ πιο μικρό από τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά, εθνικά μάλλον, συστήματα και από το Eurodac. Τι γίνεται τώρα με τη χρήση, υπό ποιου όρους θα μπορούσαν να ελεγχθούν τα δακτυλικά αυτά αποτυπώματα το 2015, ε, όπως σας είπα, ε, το ε, ΣΥΣ ε, είχε ελεγχθεί και είχαν υπάρξει 3, 3 δισεκατομμύρια χρήσεις του ΣΥΣ. Α, σίγουρα σε κάποιες περιπτώσεις θα ελεγχθούν και τα δακτυλικά αποτυπώματα. Σε κάτι αφορά, για παράδειγμα, τα προξενία, ε, σε ό,τι αφορά την έκδοση θεωρήσεων, όταν γίνεται έλεγχος από το προξενείο, ελέγχεται το σύστημα ΒΙΣ. Και ένας λόγος άρνησης χωρίς θεώρησης είναι να υπάρχει αλέρτ ε, για την είσοδο στο ΣΥΣ. Άρα είναι το θέμα αυτό των δακτυλικών αποτιμημάτων σε ό,τι αφορά το αίτημα για θεωρήσεις. Άλλο θέμα. Αναγνώριση στα σύνορα για σύνορα των χωρών των να καταφθάνουν. Δεν είναι μυστικό ότι το σύστημα εισόδου-εξόδου εντοπίζει και τα άτομα βάσει των δακτυλικών αποτυπωμάτων και εκ παραλλήλου θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αυτό για να ξεκινήσει η έρευνα στο ΣΥΣ βάσει των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Και υπάρχει και δυνατότητα που προβλέπεται επίσης σε ό,τι αφορά τα κινητά, τους κινητούς σταθμούς ή στα, αστυνομικά τμήματα, να ελέγχεται ο κόσμος στην επικράτεια των κρατών μελών. Όπως σας είπαμε, το σύστημα δεν θα λειτουργούσε σε ό,τι αφορά τα τα αδρανή, τα αποτυπώματα. για άτομα τα οποία είναι γνωστά στις αρχές σε ό,τι αφορά τη χρήση αυτών των ανδρανών αποτυπωμάτων. Θα χρησιμοποιούνταν μόνο σε περίπτωση αγνοωμένων και υπάρχουν 40 περιπτώσεις αγνοωμένων παιδιών που υπάρχουν στο ΣΥΣ. Άρα δηλαδή ή αν σε κάποιον έλεγχο αποδειχθεί ότι τα δακτυλικά αποτυπώματα σε κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο προ... προέρχεται από ένα αγνοούμενο άτομο, από ένα αγνοούμενο παιδί, τα αποτυπώματα αυτά θα μπορούσαν να προσθεθούν στην ειδοποίηση για το άτομο που έχει χαθεί. Η εφαρμογή τώρα θα ήταν αρκετά σταδιακή. Αυτή η λειτουργία, αυτή η υπηρεσία στη Γιουλίζα θα μπορούσε να αντιτεθεί σύντομα και η ακριβή διατύπωση του 22 γ δεν προβλέπει υποχρέωση για τα κρατη να χρησιμοποιήσουν αυτή τη λειτουργία, άρα δεν πιστεύουμε ότι θα ξεκινούσαν όλα τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν το σύστημα το 2017, αλλά πιστεύουμε ότι στα σταδιακά θα υπήρχε εφαρμογή. Υπάρχουν ήδη κράτη-μέλη που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα και μπορεί και κάποιοι λοιπόν να ξεκινήσουν σύντομα, κάποιοι άλλοι να καθυστερήσουν. Το επόμενο βήμα θα είναι η συνεργασία σε επίπεδο κρατών μελών, σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων για να οριστούν οι να οριστεί η ποιότητα των δακτυλικών αποτυπωμάτων και αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία, να υπάρχει η σωστή ποιότητα προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιούνται για να ζητήσει τα δακτυλικά αποτυπώματα και να οριστούν οι όροι για τον χρόνο αντίδραση, για την ποιότητα, για τις προσδοκίες, σε ποιες περιπτώσεις θα χρησιμοποιούνται. Ξεκινήσαμε τις συζητήσεις ε, σε ό,τι αφορά το Ιουλίζα και θέλουμε να εφαρμοστεί το σύστημα μέχρι το δεύτερο έμιση του έτους. και μετά να κοιτάξουμε και θέματα συγκεκριμένε εφαρμογή. Και αυτό θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2017. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για αυτές τις εξηγήσεις. Έχουμε μακρά ιστορία τεχνικών που λειτουργούν στα συστήματα SIS και σε άλλα συστήματα και μπορεί να ήταν ενδιαφέρον ίσως να δούμε αν θα λειτουργήσει και πώς μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα ώστε πράγματι το 2017 να ξεκινήσει. Ε, κάποιοι συνάδελφοι έχουν ασχοληθεί με αντίστοιχα θέματα και θέλουν να λάβουν το λόγο. Νομίζω ότι ο πρώτος που ζήτησε το λόγο ήταν ο κύριος Κοέλιο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έκθεση αυτή και να σας πω ότι είναι χρήσιμο να υπάρχουν δακτυλικά αποτυπώματα στο σύστημα για τους λόγους που ακούστηκαν φυσικά, αλλά και για δύο επιπλέον. Πρώτον, είπε εκπρόσωπος της Κομισιόν η κλοπή ταυτότητας είναι ένα από τα εγκλήματα τα οποία είναι σε αύξηση. Και επίσης για να καταπολεμήσουμε το πρόβλημα του λεγόμενου John Smith. John Smith σημαίνει ότι υπάρχει ένα πολύ συχνό όνομα τεπώνυμο και μπορεί να διώκεται κάποιος για τους λάθους λόγους. Γιατί εμείς αναζητούμε κάποιον με το ίδιο όνομα τεπώνυμο αλλά όχι το συγκεκριμένο. Η εισαγωγή λοιπόν δακτυλικών αποτυπωμάτων είναι ένας ε, καλός τρόπος να κάνουμε διάκριση μεταξύ του σωστού και του λάθους ατόμου που θέλουμε να ε, συλλάβουμε ή να βοηθήσουμε. Ένα δεύτερο το οποίο θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι στις ε, τελευταίες εκθέσεις που λάβαμε πριν από αρκετά χρόνια ένα από τα βασικά προβλήματα ήταν η ποιότητα των δακτυλικών αποτυπωμάτων τότε περίπου το 25% των δακτυλικών αποτυπωμάτων ήταν άχρηστα, γιατί ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνονταν δεν ήταν σωστός. Από την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, αντιλαμβάνομαι ότι πλέον ε, υπάρχει και η σχετική μελέτη του Κοινού Κέντρου Έρευνας που ζητά να χρησιμοποιείται το live scan, δηλαδή τα δακτυλικά αποτυπώματα να λαμβάνονται απευθεία από την οθόνη και όχι με το παλιό σύστημα με τη μελάνη που μετά έπρεπε να σαρωθεί το δακτυλικό αποτύπωμα από το χαρτί στο οποίο είχε αφήσει κάποιο το αποτυπωμά του. Αυτά τα προβλήματα λοιπόν τα οποία που διαπιστώσαμε στο παρελθόν μπορούν να βελτιωθούν τώρα σε πολύ ε, μεγάλο βαθμό. Κύριε Πρόεδρε, επίσης να πω ότι ήθελα να θίξω κάτι που δεν έχει απαραίτητα σχέση με αυτή την έκθεση, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα εμείς από πλευρά Επιτροπής ε, ΛΥΜΠΕ και πρέπει να το εξετάσει και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τα διάφορα έγγραφα. Ε, έχουμε λοιπόν ε, έγγραφα σαν αυτά ε, εδώ έχω ένα ηλεκτρονικό βιομετρικό διαβατήριο που έχει πάνω το, δακτυλικό μου αποτόπωμα και μπορεί να αποδείξω ότι πρόκειται για εμένα. Ε, δηλαδή το δακτυλικό μου αποτύπωμα είναι μέσα στο τσίπ ε, και η φωτογραφία μου. Εάν όμως είναι παραποιημένο το διαβατήριο και μπορεί να μην είναι η φωτογραφία μένα αλλά να μην είναι το σωστό όνομα. Μπορεί κάποιος να χρησιμοποιηθεί ε, να χρησιμοποιεί ένα διαβατήριο που έχει τη φωτογραφία και το δικό μου δαχτυλικό αποτύπωμα, αλλά άλλο όνομα τεπώνομο. Θα πρέπει λοιπόν να διευκρινίσουμε πώς μπορούμε να ε, εγκρίνουμε την έκδοση αυτών των συγκεκριμένων διαβατηρίων. Δεν μπορούμε να νομοθετήσουμε, ε, αλλά για να εμπιστευόμαστε αυτά τα έγγραφα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό πώς εκδίδουν τα συγκεκριμένα έγγραφα τα κράτη-μέλη, πώς επαληθεύουν ότι όντως πρόκειται για το σωστό ιδιοκτήτη του εγγράφου. Σίγουρα θα πρέπει να ενισχύσουμε την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και παρά το γεγονό ότι γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να νομοθετήσουμε επί του ζητήματο, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα σε πολιτικό επίπεδο. Εάν θέλουμε να εμπιστευόμαστε τέτοια έγγραφα, πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι η διαδικασία έκδοσή του είναι ε, με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ ως ε, εισηγητής για τα θέματα αυτά ξέρετε όλες αυτές τις λεπτομέρειες πολύ καλύτερα από μένα, αλλά το πόσο ασφαλή είναι αυτά τα έγγραφα και πόσο εύκολα μπορεί κάποιος ε, να τα παραποιήσει είναι σίγουρα ιδιαίτερα σημαντικό και θα ήθελα να τονίσω ότι πέραν ε, του θέματος της ποιότητας των δακτυλικών αποτυπωμάτων που λαμβάνονται υπάρχει και ένα θέμα που αφορά τα δακτυλικά αποτυπώματα με τους ανήλικους ε, που μπορεί να αλλάξουν δακτυλικό αποτύπωμα όταν ενηλικιωθούν. Ο κύριος Ντεπρέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Απλά μίλαγα με τη Σοφή και είχα αφιερωθεί εντελώς. Είχα αφιερωθεί την προσοχή μου στη Σοφή. Αλλά τώρα πιο σοβαρά. Να πω ότι με ικανοποίηση στα συμπεράσματα της έκθεσης διαβάζω ότι η τεχνολογία ταυτοποίησης μέσω των δακτυλικών αποτυπωμάτων ε, είναι διαθέσιμη και έτοιμη να συμπεριληφθεί στο ΣΥΣ 2 Όσοι θυμάστε τις δυσκολίες εγκατάστασης του ΣΥΣ2 και τις μεγάλες και πολλές εκπλήξεις που αντιμετωπίσαμε, είναι εξαιρετικό το νέο. Αυτό οφείλω να το επισημάνω. Τώρα, έχω αρκετές ερωτήσεις. Ε, στην έκθεσή σας, ε, κυρία μου, λέτε πίσω ότι εξολογείτε την τεχνική ικανότητα ε, για τη γρήγορη ε, εξέταση των δακτυλικών αποτυπωμάτων, ε, φαντάζομαι κατά τη διέλευση των συνόρων. Μιλάμε για δευτερόλεπτα υποθέτω. Ισχύει αυτό για την επαλήθευση. Σε ό,τι αφορά τώρα τη φάση της εγκατάστασης για τα εφή σύνορα μιλώ, τι θέση θα έχει αυτό. Επίσης είπατε ότι αυτό είναι το πιο ευφυές σύστημα ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ασφάλεια. Αν έχω σωστές πληροφορίες, αυτό το σύστημα έχει 800.000 ε, στοιχεία για άτομα, για πρόσωπα, αλλά μόνο 90.000 δακτυλικά αποτυπώματα. Και αυτό εξηγείται αν λάβουμε υπόψη ότι το άρθρο 23 παράγραφος 2 της απόφασης Τζάι του 2007 λέει ότι τα ψηφιακά αποτυπώματα μπορούν να προσθεθούν αν ένα κράτος μέλος έχει στη διάθεσή του τέτοιου είδους αποτυπώματα. Το... Τα πρώτα κράτη-μέλη δεν τα είχαν. Γιατί δεν λέτε ότι ο κανόνας είναι ότι όταν ένα κράτος μέλος που δεν είναι το κράτος που ζήτησε την έχει ψηφιακά αποτυπώματα... να τα συμπεριλάβει. ώστε αυτό τελικά να γίνει κανόνας. Δεν ξέρω πώς έχω, δεν έχω καταλάβει καλά. Λέτε κάποια πράγματα που κυκλοφορούν παράνομα και το κείμενο θεώρησε το άρθρο 7 του κώδικα Σέγγεν που καθιστά τους του ελέγχου ε, στα σημεία εισόδου-εξόδου του χώρου Σέγγεν προβλέπει ότι τα βιομετρικά στοιχεία των διαβατηρίων και των ταξιδιωτικών εγγράφων που χορηγούνται πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο επαλήθευσης. Καλά τα διαβάζω. Υπάρχουν και πολλές ε, περιπτώσεις όπου πολίτες της Ένωσης που θα ελέγχονται ε, συστηματικά δεν χρειάζονται διαβατήριο ή κάποιο άλλο συγκεκριμένο ταξιδιωτικό έγγραφο για να μεταβούν σε ορισμένες χώρες, όπως για παράδειγμα πάνω από το Βέλγιο στην Ιρλανδία ή στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στο Μαρόκο ή στην Τινησία. Δεν χρειάζονται διαβατήριο. Αρκεί η ταυτότητα. Το ερώτημά μου είναι, στη λογική παράταση που θέλουμε να κάνουμε με το ΣΥΣ, μήπως θα έπρεπε για τις ταυτότητες, να προσπαθήσουμε να ομοιογενοποιήσουμε τους κανόνες βάσει των οποίων τα βιομετρικά στοιχεία που περιλαμβάνουν θα πρέπει να τηρούν κάποιους κοινού κανόνες. Δεν είναι αντικείμενο της πάθος απόφασης, αλλά νομίζω ότι είναι φυσική επέκταση το τι θέλουμε να κάνουμε σήμερα. Γιατί αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ένα μέσο για να λέγουμε συστηματικά όλους τους επιβάτες, αλλά έχουμε μόνο διαβατήρια και ταξιδιτικά έγγραφα, αυτοί που μπορούν να κυκλοφορούν μόνο με ταυτότητα δεν ελέγχονται. Αποτελεσματικά τουλάχιστον. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Έχω κι άλλα. Δεν είναι όμω τόσο επίγοντα, άρα μένω σε αυτά. Προς το παρόν ευχαριστώ. Προς ευχαριστώ πολύ κύριε Ντεπρέ. Πολλές είναι οι ερωτήσεις σε σχέση με τις τεχνικές δυνατότητες, το ερώτημα πόσο ασφαλή είναι τα αποτυπώματα, το θέμα των ασφαλών εγγράφων και υπάρχει και το ερώτημα κατά πόσον όλα τα κρατη οι αρχές στα κράτη-μέλη είναι σε θέση να εξασφαλίσουν ότι αν εγώ πάω και πω ότι θέλω ένα νέο διαβατήριο και με λένε Ματίνα Μίλλερ, που δεν ισχύει αυτό, θα το ξέρει η αρχή αρμόδια ότι δεν είναι η εκδούσα αρχή. Άρα και αυτό είναι ένα ερώτημα και έπειτα. Το σύστημα τελικά πόσο γρήγορο είναι. Πόσο θα είναι στην πράξη. Αυτά είναι τα ερώτημα. Δεν βλέπω να θέλει το λόγο κάποιο άλλο συνάδελφο, οπότε και ο Γέννησαν θα μπορούσε ενδεχομένω να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι ευγνώμων για τις ερωτήσεις. Σε ό,τι τεχνικό σκέλος θα δώσω αργότερα το λόγο στον συνάδελφό μου, τον Ρίτσαρντ, ο οποίος μπορεί να απαντήσει τα πολυτεχνικά ερωτήματα και εγώ θα ήθελα να απαντήσω ορισμένα από άλλα, ορισμένα άλλα από τα ζητήματα που θέσατε. Ο κύριος Κοέλιο είπε, ποιότητα των αποτυπωμάτων που είναι στο σύστημα δεν είναι ομοιόμορφη. προβλέπεται το πρώτο 2000 και είναι και στο εγχειρίδιο, άρα είναι δεσμευτικό, όμως τα κράτη-μέλη έχουν φακέλους JPEG ή e PDF που κατεβάζουν ε, και ανεβάζουν μετά στο σύστημα. Όλα λοιπόν τα αρχεία τα οποία δεν ε, θα συμμορφούνται προς το πρότυπο το νέο θα απορρίπτονται από το σύστημα. Εμείς θέλουμε λοιπόν να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου αυτόματα μέσα στο νέο σύστημα. Δηλαδή να υπάρχει ένα τσέκερ, ένα, ε, ένα λογισμικό που θα ελέγχει ποια είναι τα αρχεία τα οποία είναι συμβατά με το νέο πρότυπο και ποια δεν είναι. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στα αποτυπώματα των ανηλίκων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα. Στο Eurodac ε, από τα 14 και μετά παίρνουν δακτυλικά αποτυπώματα από ανηλίκους. Δεν υπάρχει τώρα εδώ ένα όριο γιατί είναι θέμα εθνικής νομοθεσίας αλλά είδαμε ε, από μια τελευταία έκθεση GRC ότι από τα έξι μπορούν να ληφθούν αποτυπώματα ε, από ε, άτομα ανήλικα με αξιόπιστο τρόπο και λαμβάνονται υπόψη το πώς μεγαλώνοντας μπορεί να αλλάζουν τα δεκτικά αποτυπώματα και να γίνεται μια σύγκριση μετά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους ασυνόδευτους ανήλικους, πριν από δύο χρόνια η Ιταλία παρατήρησε ότι φτάνουν ανήλικοι που καταγράφονται, καταχωρίζονται στο τελικό σύστημα, χωρίς δακτυλικά αποτυπώματα, αλλά επειδή δεν θέλουν να παραμείνουν στην Ιταλία, δεν καταθέτουν αίτηση ασύλου, καταγράφονται ως παράτυποι μετανάστες. Οι Ιταλικές αρχές τις, τους ανθρώπους αυτούς καταγράφουν ε, στο ΣΥΣ, αλλά υπάρχει μόνο στο Λίμα ε, το Όνομα, τεπώνυμο και ημερομηνία γέννηση. Και αυτά τα παιδιά λοιπόν ε, περιπλανούνται από εδώ και από εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν υπάρχει σύστημα που θα μπορούσε να τα ταυτοποιήσει. Αν επομένως ε, συλληφθούν και πούν ένα άλλο όνομα σε ένα άλλο κράτος μέλος, δεν μπορεί το σύστημα να τα βρει. Στο σύστημα Eurodac καταγράφοντας παράτυποι μετανάστες μένα, αλλά δεν υπάρχει νομικά το ενδεχόμενο να ληφθούν τα δακτυλικά τους αποτυπώματα στο Eurodac και αυτό είναι ένα κενό, είναι ένα πρόβλημα. Το αναγνωρίσαμε και με βάση το Ιταλικό project ε, θεωρήσαμε ότι το όριο ηλικίας για τους αρισινόδευτους ανηλίκους θα πρέπει να είναι κατώτερο για την καταχώρηση και αν ε, καταγράφονται με βάση κάποιο δακτυλικό αποτύπωμα στο ΣΥΣ, ε, σίγουρα θα μπορούσε αυτό να γίνεται πριν την ηλικία των 14. Ο μέσος όρος άλλωστε των ανηλίκων, των ασυνόδευτων ανηλίκων μειώνεται από γίνει γύρω στα 12 με 14. Για το χρόνο απόκρισης, response time, εξαρτάται από την κατάσταση στα σύνορα. Τώρα με το ΒΕΕΣ αυτό που είδαμε είναι ότι το σύστημα μπορεί να δίνει απάντηση μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Και αυτό εξαρτάται βέβαια από την εθνική εφαρμογή και το εύρος του δικτύου, την ευρυζωνικότητα του δικτύου. Επαναλαμβάνω, εξαρτάται από την εθνική εφαρμογή. Στα αεροδρόμια, στα σύνορα, σίγουρα θα υπάρχει απέτηση να είναι σε δευτερόλεπτο χρόνος απόκρισης. Το συζητήσαμε πάντως αυτό, είχαμε και το feedback από τα κράτη-μέλη. Δέκα δευτερόλεπτα θεωρούν ότι είναι πολύ μεγάλο το χρονικό αυτό. Διάστημα πρέπει να μειωθεί, αλλά αν κάποιου ληφθούν σε ένα αστυνομικό με τα τακτυλικά του αποτυπώματα, αν ο χρόνο απόκριση είναι λίγα δευτερόλεπτα, δεν είναι και τόσο κακό. Ξερτάται πάντα από τη συγκεκριμένη περίπτωση για το χρόνο απόκριση πόσο μικρό θα πρέπει να είναι. Επίσης για το ΣΥΣ μέσα σε δύο δευτερόλεπτα έχουμε απόκριση. για τις ταυτότητες και τα λοιπά. Θα δώσω το λόγο στον Ρίτσαρτ από την δική μου τη μονάδα που ασχολείται με την ασφάλεια των εγγράφων. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να απαντήσω λοιπόν στην ερώτηση του κυρίου Κοέλιο. Η ακρίβεια ενός αυτοματοποιημένου συστήματος δακτυλικών αποτυπωμάτων εξαρτάται ακριβώς από την ποιότητα των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Στην πρώτη περίοδο του συστήματος VIS, όταν έγιναν πάρα πολλές συζητήσεις στη συγκεκριμένη ομάδα, αποφασίστηκε να γίνεται ένας έλεγχος ποιότητος στο σημείο καταχώρησης, που ε, σήμαινε ότι αν τα, η ποιότητα των ε, συστήματος VIS ε, ή τα δακτυλικά αποτυπώματα είναι πάρα πολύ χαμηλά ώστε να μην έχουμε εξαιρετική ακρίβεια, τότε δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι τότε τα δακτυλικά αποτυπώματα λαμβάνονταν από άτομα τα οποία δεν ήταν τόσο ε, καλά ε, εξειδικευμένα στο να λαμβάνουν δακτυλικά αποτυπώματα. Προξερικές αρχές, για παράδειγμα, του Υπουργείου Εξωτερικών Υποθέσεων. Ελπίζουμε αυτή τη φορά να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα είναι πάρα πολύ καλοί γνώστες της λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων. Το Κοινό Κέντρο Έρευνας επισκέπτηκε ε, διάφορα κράτη-μέλη και εξέτασε την ποιότητα των δακτυλικών αποτυπωμάτων ε, στο σύστημα άφηση της αστυνομίας και διαπίστωσαν με έκπληξη ότι η ποιότητα των δακτυλικών αποτυπωμάτων είναι ιδιαίτερα υψηλή. Όπως είπε και ο κύριος Κοέλιο, ακολουθήσαμε την ίδια ε, κατεύθυνση με το VIS. Άρα τα δακτυλικά αποτυπώματα θα λαμβάνονται με εξοπλισμό ζωντανής ε, σάρωσης. Ε, η παλιά εποχή του Hollywood με δακτυλικά αποτυπώματα με μελάνι έχει περάσει προπολού. Όσον αφορά τώρα τα έγγραφα, τα βιομετρικά, ε, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πόσα προγράμματα έχουν υπάρξει στους πρόσφατους μήνες. Παραδείγματος χάρη έρευνα βάσει του Fidelity μας έδειξαν ότι ε, πρέπει κάτι να γίνει. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή είναι πολύ περιορισμένη η πόρη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι από αυτό. Από πολιτική σκοπιά ίσως θα μπορούσε να αλλάξει τίποτα ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση δεν είναι μόνο τα βασικά έγγραφα αναγνώρισης ταυτότητας, διαβατήρια κλπ, αλλά είναι ε, παραμόρφωση της ε, εικόνας ενός ανθρώπου. Δύο φωτογραφίες δύο διαφορετικών ατόμων συνδυάζονται σε μία. Πρόκειται για τους δύο ανθρώπους που χρησιμοποιούν το ίδιο διαβατήριο για να περάσουν τα σύνορα. Η ηλικία σαφώς επηρεάζει τα δακτυλικά αποτυπώματα, τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματα ο κύριος Κοέλιο γιατί η χώρα του συμμετείχε σε έρευνα που έγινε επί του ζητήματος και η έρευνα σαφώς καταδεικνύει ότι αν εφαρμοστούν οι βέλτιστες πρακτικές, ε, τα δακτυλικά αποτυπώματα μπορούν να χρησιμοποιούνται από την ηλικία των 6 ετών και μετά οι αλλαγές ε, καθώς μεγαλώνει ένα παιδί είναι τόσο περιορισμένες ε, που δεν επηρεάζεται το δακτυλικό τους αποτύπωμα. Όσον αφορά το, την ερώτηση του κυρίου Ντεπρέ, η ταχύα αναζήτηση θα εξαρτάται καταρχάς από το πώς ε, κονδύλια δαπανούνται στο σύστημα ε, το οποίο ε, θα κάνει διασταύρωση δακτυλικών αποτυπωμάτων. Δεύτερον, μας ενδιαφέρει η ποιότητα και τρίτον, πάρα πολύ σημαντικό, ε, πόσα αρχεία θα πρέπει να εξετάσει το σύστημα. Το VIS ήταν κατασκευασμένο για να εξετάζει 70 εκατομμύρια δακτυλικά αποτυπώματα μέσα σε λίγα λεπτά. Το σύστημα αυτό πλέον είναι λίγο παλιό, τα πράγματα έχουν εξελιχθεί. Το SIS κατά πάσα πιθανότητα θα ε, εξετάζει ένα εκατομμύριο δακτυλικά αποτυπώματα το πολύ. Ε, εξετάζουμε το σύστημα με χώρες που σε όλη την Ιφίλιο έχουν χρησιμοποιήσει αντίστοιχα συστήματα. Ε, μπορεί να γίνεται αναζήτηση σε 2-3 δευτερόλεπτα ενός εκατομμυρίου δακτυλικών αποτυπωμάτων εάν τα δακτυλικά αποτυπώματα λαμβάνονται για τα FEE e σύνορα, για υπηκόους τρίτων χωρών ε, στα σημεία εισόδου-εξόδου ε, σε ένα σύστημα, τότε μπορούμε να έχουμε μια αντίστοιχη λειτουργία και για ένα σύστημα εισόδου-εξόδου και, και για ένα σύστημα πληροφοριών Schengen αν κάποιος ε, στο σημείο εισόδου δίνει τα δακτυλικά του αποτυπώματα, τότε μπορούμε κάλλιστα να κάνουμε αναζήτηση στο σύστημα SIS ε, για να δούμε αν υπάρχει ε, άρνηση εισόδου για το συγκεκριμένο άτομο. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην δημιουργήσουμε ένα αμάλγαμα, αν μου επιτρέπετε η χρήση του όρου, μεταξύ των ε, ταξιδιωτικών εγγράφων ε, και του συστήματος ε, βιομετρικής επαλήθευσης και του συστήματος βιομετρικής επαλήθευσης του SIS. Όλοι κατά πάσα πιθανότητα έχουμε ηλεκτρονικά διαβατήρια με τη φωτογραφία μας και τα δακτυλικά μας αποτυπώματα. Η πρόταση τροποποίησης του SIS λέει συγκεκριμένα ότι θα πρέπει τουλάχιστον στο σημείο εισόδου των συνόρων να είμαστε βέβαιοι ότι το έγγραφο ανήκει σε αυτόν που το φέρει. Ε, πρέπει λοιπόν να γίνεται μια επαλήθευση ε, από ένα συνοριοφύλακα ή μέσω ενό μηχανήματο θα συγκρίνεται με τη φωτογραφία που περιλαμβάνεται στο τσίπ. Αυτό στην ουσία έχει ελάχιστη σχέση με μια πιθανή αναζήτηση δαχτυλικών αποτυπωμάτων στο SIS. Εάν ε, γίνεται ένα έλεγχο στα σύνορα βάσει της ε, φωτογραφία σα. και για οποιοδήποτε λόγο ο συνοριοφύλακα έχει λόγο να πιστεύει ότι μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, μπορούμε να ε, κάνουμε ένα δεύτερο έλεγχο και εκεί ε, να επισέλθουμε σε όλες τις μορφές ε, περαιτέρω ελέγχων. Αλλά η πρόταση για τις αλλαγές στο SIS αφορά τον αρχικό πρώτο έλεγχο με βάση το ταξιδιωτικό έγγραφο. Πολλοί αναφέρθηκαν στην ομογενοποίηση των ε, κοινών ε, ε, χαρακτηριστικών ασφαλείας για τις ταυτότητες. Είναι γνωστό τη πάση ότι αυτή τη στιγμή οι πολίτες μπορεί να χρησιμοποιήσουν την ταυτότητά τους όχι μόνο για να φύγουν από το χώρο Σέγγεν αλλά και να επανέλθουν, αλλά μπορούν να επισκεφθούν και τρίτες χώρες. Η Τινησία, για παράδειγμα, αναφέρθηκε. Αν όμως έχω ε, μια ταυτότητα σε χαρτί με ελάχιστα χαρακτηριστικά ασφαλείας και ε, από την άλλη έχω και ένα διαβατήριο τελευταίας γενιάς με ε, δακτυλικά αποτυπώματα και τα πάντα σε, που να περιλαμβάνονται μέσα, σίγουρα κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Προσπαθούμε λοιπόν να εναρμονίσουμε λίγο τη διαδικασία και υπάρχει σχετική μελέτη. Αυτά σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε λέει η Πρόεδρος. Ε, ήταν πραγματικά πολύ χρήσιμη η συζήτηση αυτή σήμερα και θα διοργανωθούν ασφαλώς ε, και άλλες συζητήσεις. Δεν υπάρχει ακόμα σχετικό χρονοδιάγραμμα. Θα ξεκινήσουμε τις εργασίες μας για την κατάρτιση σχετικού ψηφίσματος. Θα παρουσιάσουμε τις απόψεις μας για την ε, πρόταση αυτή. Θα υπάρξει και επιπρόσθετη συζήτηση για κάποια θέματα τα οποία αναφέραμε σε ό,τι αφορά τα ευφυή σύνορα και το σύστημα αξιολόγησης του ΒΙΣ ε, έχω κάποιες αμφιβολίες για το κατά πόσον η χρήση όλων των αποτυπωμάτων ανα πάσα στιγμή θα βοηθήσει. Αλλά αυτή είναι μια συζήτηση ε, επί της ουσίας ε, θεμελιώδης, γιατί στη Γερμανία μπορεί κανείς να βάλει τα δακτυλικά του αποτυπώματα στην ταυτότητα και ως τώρα το αρνούμε εγώ προσωπικά γιατί δεν βλέπω τι χρησιμότητα έχει ακριβώς. Το θέμα είναι λοιπόν αν υπάρχει, κατά πόσον είναι ασφαλής. Θα υπάρχει πραγματική εγγύηση ότι θα υπάρχει σύνδεση με το άτομο με το οποίο θα πρέπει να συνδέεται. Υπάρχει επίσης ε, δυνατότητα να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα ε, χακαριστεί, δεν θα έχει κάποιος άλλος πρόσβαση σε αυτό το στοιχείο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν για τη συζήτηση αυτή και τώρα θα πρέπει να περάσουμε στην ψηφοφορία. Να υπενθυμίσω σε όλους ότι θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε την κάρτα ψηφοφορία σας. Όσοι δεν το έχουν, δεν την έχουν μαζί τους, έχουν λίγο χρόνο. Γιατί η ψηφοφορία θα ξεκινούσε στις 6 και 20. Και δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία και σε 10 λεπτά να, μάλλον να μην μπορέσουν να ψηφίσουν οι συνάδελφοι. Έχετε λοιπόν λίγα λεπτά παραπάνω και θα ήθελα 6 και 18 να είστε στην αίθουσα για να ξεκινήσει η ψηφοφορία. Συγγνώμη και σας ευχαριστώ. So, okay, it's now 6.20. Λοιπόν, 6 και 21 είναι. Σας δίνω ένα λεπτό ακόμα για να είμαστε βέβαιοι ότι έχετε όλοι τις κάρτες σας και θα ψηφίσουμε. εφαρμογή της οδηγίας του Συμβουλίου κλπ. κλπ. που καθορίζει ένα γενικό πλαίσιο για ίση μεταχείριση στην απασχόληση η οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση. Η συγγήτρια ήταν η Χέλγα Στίβενς, δεν ξέρω αν θέλει να πει δυο λόγια. Okay, so we can... Ωραία, μπορούμε να περάσουμε απευθεία στην ψηφοφορία. Θα γίνει ηλεκτρονικά. Τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορριπτεται, σαφέστατα. Τώρα, τροπολογία 2, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3 και τροπολογία 4 καταπίπτουν. επιβαστική τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρινέται. Πάμε απευθείας λοιπόν στην τροπολογία 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Οι επόμενες λοιπόν τροπολογίες καταπίπτουν και πάμε στη συμβαστική τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 15. Άρχεται η ψηφοφορία. πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 23, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε το κείμενο ως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται σαφέστατα συγχαρητήρια στην εισηγήτρια και καλό σας βράδυ. Πέρασε της συνεδρίασης.